Finger. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Sitzung unseres Καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής μας ε, την καινούργια χρονιά σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες και Βεβαίως είμαστε στο τέλος της θητείας μας ε, αλλά έχουμε μέχρι το τέλος Μαΐου να δουλέψουμε όπως βλέπετε όπως βλέπετε ε, είμαστε στο καινούριο κτίριο του Κοινοβουλίου με το με τις μοντέρνες αίθουσες ε, ε, και αύριο θα έχουμε ε, θα είμαστε και στην θα βγούμε και στην τηλεόραση στο διαδίκτυο μάλλον η κάμερα θα παρακολουθεί το μικρόφωνο οπότε έχετε το υπόψη σας Λοιπόν, σημείο 1, ημερήσια διάταξη, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, πρώτο θέμα που μας σας δόθηκε έγκαιρα. Τώρα, ο Φελίπε Γκοντζάλες ε, πρέπει να γυρίσει στη Μαδρίτη και έχει ένα αεροπλάνο για τη Μαδρίτη και το Οπότε θέλουμε, πρέπει να αλλάξουμε νομίζω λίγο την ε, ημερήσια διάταξη και θα συζητούμε βέβαια όταν έρθει ο κύριος Κονζάλες μάλλον την έκθεση Elmar Brock εάν ε, δεν έχουμε τελειώσει τη συζήτηση θα πρέπει να διακόψουμε τη συζήτηση για να ε, ανταλλάξουμε απόψη με τον κύριο Γκονζάλες τώρα το σημείο 9 της σας διάταξης. Ο κύριος Δημητρίου αύριο πρέπει να φύγει για Κύπρο και ζήτησε αν είναι δυνατόν αύριο το πρωί νωρίς η έκθεσή του να ψηφιστεί για να μπορέσει να φύγει. Θα ήθελα τώρα να ε, καλωσορίσω καινούριου συναδέλφους που όμως δεν βλέπω να είναι εδώ. Βλέπω απλώς τον κύριο Κάστλερ που αντικαθιστά τον κύριο Φρίντριχ είναι ο μόνος καινούριο που είναι εδώ ε, οι άλλοι δεν είναι εδώ τώρα για το περίφημο web streaming αυτή την, ε, το ίντερνετ που σας λέω ε, στο οποίο θα βγούμε αύριο τα είπα προχωρώ στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης Mitteilung des Vorsitzenden. Die Koordinatoren haben zweimal. Λοιπόν, οι συντονιστές ε, συναντήθηκαν 17 Δεκεμβρίου και 14 Ιανουαρίου και ε, το ΙΣ 15 και πρότειναν ε, οι εκθέσεις Λάινεν, Μπροκ και να συζητηθούν ε, επιγόντως είναι για την συνθήκη της Λισαβόνας ε, σχετικές οι εκθέσεις αυτές για να μπορέσουν να εγκριθούν να περάσουν στην Ολομέλεια του Απριλίου τώρα βέβαια το Συμβούλιο τι θα κάνει δεν ξέρουμε αυτό αφορά κύρια την έκθεση Μπροκ τώρα για την έκθεση Κόρβετ σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του κανονισμού ε, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών ε, επεκτείνεται, παρατείνεται μέχρι τις 10 ε, Φεβρουαρίου Αυτά για τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Τώρα για τα πρακτικά. 3η και 4η Νοεμβρίου, 17η Νοεμβρίου και 1η και 2η Δεκεμβρίου. Εάν μέχρι το τέλο τη συνεδρία δεν πείτε τίποτα, θα τα θεωρήσω αυτά τα πρακτικά εγκεκριμένα. Ε, προχωρώ στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήδη ε, από την περασμένη φορά ξεκινήσαμε την συζήτηση αυτή του χαπί του είχα πει του κυρίου Μπρόκ ότι θα έρθει 4 παρα 10 ο, ο κύριος Γκονζάλες ε, δεν ξέρω τώρα ε, τι θέλεις θέλεις να πάρεις το λόγο Αλμαρ ή να μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση Ωραία δεν θέλει ο κύριος Μπροκ το λόγο Οπότε κερδίζουμε χρόνο Την έκθεση του μεταξύ την έχετε πάρει σε όλες τις γλώσσες Οπότε άρχεται η συζήτηση Αγαπητοί συνάδελφοι από πλευράς μου εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι θεωρώ αποδίδω τεράστια σημασία στις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Η κοινοβουλευτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί ε, σε τελευταία ανάλυση πρέπει να δουλεύουμε για τους πολίτες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία ε, χρόνια από την εποχή της συνέλευσης ε, έχουν ενισχυθεί η σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια ε, γίνονται όλο και πιο πολλές συναντήσεις και επαφές και στα πλαίσια της ΚΟΖΑΚ ε, και πολλά ακόμη και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Ο διάλογος αυτός είναι και απαραίτητος για να ε, ε, διαδώσουμε αν, θες, αν θέλετε τις γνώσεις για την Ευρώπη ε, αλλά επίσης ο διάλογος αυτός βοηθάει στο να αρθούν ενδεχομένως παρεξηγήσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας τι να σας πω για όλα τα θέματα ε, και θέματα μεγάλα κιόλα που συζητούνται και σε παγκόσμιο επίπεδο τι να σας πω ε, αλλαγή του κλίματος προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Λοιπόν ευχαριστώ τον Έλμαρ Μπροκ για την έκθεσή του ε, βλέπω πια γραμμή χαράσει ο κύριος Μπροκ ε, στην έκθεσή του φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν το λόγο ε, χαιρετώ τον κύριο Λένε, ε, τον καλωσορίζω, είναι νέος στην Επιτροπή μας. Εύχομαι καλή συνεργασία. Hm? Α, έχουμε και γενέθλια. Ο Μέντες Τεβίγκο έχει γενέθλια σήμερα και για την μέρα των γενεθλίων του έρχεται στις Βρυξέλλες να συζητήσει στην Επιτροπή. Χρόνια πολλά. So, ich, ε, Λοιπόν, τώρα για, εγώ προσωπικά για την έκθεση Elmar Brock θα ήθελα να πω το εξής. Στο σημείο 2 αναφέρονται οι διάφορες μορφές ε, σχέσεων αλλά δεν αναφέρεται η γενική ε, δεν αναφέρονται οι μεγάλες ε, κοινοβουλευτικές συνελεύσεις οι ΑΣΥΣ που κάνουμε δύο φορές το χρόνο είναι το Interparliamentary Forum αυτό που λέμε αυτό λείπει από εδώ μετά στο 18 ε, αναφέρεται η Κόζακ, ο εκπρόσωπος μας στην Κόζακ είναι ο Κόρμπετ. Μάλλον, ε, μέχρι τώρα εκπροσωπούμεθα από δύο, από τον πρόεδρο της ΑΦΚΟ και άλλους ε, ε, και επειδή και τα Εθνικά Κοινοβουλία έχουν έξι εκπροσώπους και εμείς έχουμε έξι εκπροσώπους εκεί αλλά η ομάδα για τη μεταρρύθμιση της Dagmarot Berend ε, προτείνει αλλαγές για καλύτερο συντονισμό και τα λοιπά και γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε και εμείς μήπως η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών πρέπει να εμπλακεί με την ΚΟΖΑΚ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, να φτιάξουμε έτσι μια ομάδα ε, αλλιώτικη από τη μέχρι τώρα για τη συμμετοχή μας στην Κόζακ. Στο 19 ε, αναφέρεται εδώ συστηματικότερη παρακολούθηση του διαλόγου μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Επιτροπής Πρωτοβουλία Μπαρόζο στα γερμανικά αντί για παρακολούθηση αναφέρεται control δεν είναι σωστή η λέξη control στα γερμανικά ε, στα αγγλικά λέγεται monitoring οπότε νομίζω ότι και στα γερμανικά πρέπει να βρεθεί μια λέξη για την παρακολούθηση διότι δεν πρόκειται να ελέγξουμε τίποτα εκεί τώρα παρακάτω λέγεται ότι το κοινοβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να οριστεί ο μελλοντικός ρόλος της ΚΟΖΑΚ. Αυτό δεν είναι αρκετά σαφές κατ' με γιατί στον κανονισμό της ΚΟΖΑΚ και στο πρωτόκολλο της συνθήκης του Άμστερνταμ και στη νέα συνθήκη ορίζεται σαφώς ο ρόλος της ΚΟΖΑΚ. Ε, τέσσερα χρόνια ολόκληρα μεταρρυθμιζόταν αν θέλετε η Κόζακ πολύ έντονες και ζωηρές και αμφιλεγόμενες συζητήσεις οπότε νομίζω ότι ο ρόλος της Κόζακ είναι δεδομένος ε, Ίσως θα πρέπει να μιλούμε εδώ για τον πολιτικό ρόλο της Κόζακ ε, και στο τέλος του, της ε, παραγράφου 15 λέ, αναφέρεται ε, πάλι για την Κόζακ ο, επικεντρώνονται λέει ο διάλογος πρέπει να επικεντρώνεται σε νομοθετικές δραστηριότητες για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας λέει εδώ Μα έχω την εντύπωση ότι υπήρχε συνένεση πως η Κόζακ θα πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση για την ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω ε, επιχειρείται τεχνητός περιορισμός του ρόλου της Κόζακ θέλουμε κάτι τέτοιο εγώ πραγματικά παρακολούθησα την όλη διαδικασία μεταρρύθμισης της Κόζακ και σας λέω ότι τα πράγματα είναι σαφή δεν ε, μπορούμε να τα αμφισβητούμε εδώ Αυτά, αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις τώρα ζήτησε το λόγο κυρία Κραπόφσκα παρακαλώ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω γενικά για την έκθεση του κύριου Μπρόκ. Σε πολλές ευκαιρίες συζητήσαμε τις επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είχαμε τονίσει πολλές φορές την σημασία των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά αυτό που μου αρέσει κυρίως στην έκθεση είναι το εξής, ότι λέει πως ε, ναι, εν τέλει καθησυχάσαμε τα εθνικά κοινοβούλια ως προς την θεωρητική, τέλο πάντων την υποτιθέμενη βούλησή μας να περιορίσουμε τις αρμοδιότητές τους. Δείξαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη ταυτόχρονα αφήνοντας κάποια θέματα να ρηθούν από τις αμοιβαίες επαφές μας. Η συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν είναι η μόνη ε, διέξοδος. Υπάρχουν και οι σχέσεις μεταξύ βουλευτών και ευρωβουλευτών. Ξέρω ότι η έκθεση το τονίζει αυτό και ε, μάλλον η έκθεση δεν τονίζει αυτό γιατί ασχολείται με τις επίσημε δομέ συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάντων. Ωστόσο, ο συντονισμό τη θεσμική αυτή συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται και σε καλέ προσωπικέ σχέσει μεταξύ των βουλευτών που έχουν εκλεγεί στα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν άλλα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών που τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Συχνά ωστόσο προβλήματα, τα προβλήματα αυτά έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και δεν είναι αναγκαίο να μπορεί πάντα ένας εθνικός βουλευτής να τα λύσει. Ούτε από την άλλη μεριά ένας ευρωβουλευτής μπορεί να λύσει τα προβλήματα που του θέτουν οι πολίτες. Μπορεί η λύση του προβλήματος να πατάει και σε ευρωπαϊκά και σε εθνικά ζητήματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι στενότερες σχέσεις μεταξύ βουλευτών και ευρωβουλευτών στις περιφέρειες και τα κράτη μας επιτρέπουν καλύτερη εφαρμογή των συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω για την έκθεση Μπροκ. Καταρχήν, την ανάγκη να εκμεταλλευτεί η πολιτική την τεχνολογία. Οι σχέσεις μεταξύ εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν και μια συζήτηση για την ανάγκη μεγαλύτερης προσέγγισης του κέντρου λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των περιφερειών. Τούτο μπορεί να υλοποιηθεί με μορφές προσέγγισης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πώς μπορεί τούτο να γίνει χρησιμοποιώντας περισσότερο το σύστημα της βίντεο για να οργανώνουμε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στα Εθνικά Κοινοβούλια, στο εσωτερικό των Εθνικών Κοινοβουλίων, για να επιτρέπουμε να επικοινωνεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κάποιο εθνικό κοινοβούλιο που συζητά ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτό θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί. Σε κάποιες περιπτώσεις και για κάποια θέματα που μπορούμε να αποφασίσουμε έτσι οθολογικά θα μπορούσαμε να έχουμε θετικές συνέπειες. Θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών. Θα είχε ταυτόχρονα θα επέτρεπε την θέσπιση ημερησίων διατάξεων που θα ήταν πιο κοντά η μία με την άλλη και θα επέτρεπε στο, στην κοινή γνώμη της Ευρώπης να παρακολουθήσει καλύτερα τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Επιπλέον θα προσέφερε και μία ε, καλύτερη αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών θεμάτων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα μέσα. Όταν Αν προσεγγίζαμε, φέραμε κοντά τις τα ζητήματα που απασχολούν το τα εθνικά κοινοβούλια με αυτά του Ευρωπαϊκού θα μπορούσαν να διευκολύνουν αυτή τη φυσική προσέγγιση. Εγώ δεν λέω να μεταφέρουμε τις δραστηριότητες των Βρυξελών ή του Στρασβούργου στο εθνικό πλαίσιο. Αλλά σε κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία όλες οι, όλα τα πολιτικά μοντέλα έχουν ε, μπερδευτεί, το να μην εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία που, μια τεχνολογία που έχει διεθνές ε, αντίκρισμα και να παραμένουμε σε δομές λειτουργίας του περασμένου αιώνα είναι παράλογο. Θα έπρεπε λοιπόν από καιρούς καιρών ε, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές του κοινοβουλίου μας θα έπρεπε να μπορούν να συναντηθούν με εθνικά κοινοβούλια μέσω βίντεο διασκέψεων. Αυτό θα είχε θετικές συνέπειες για τη βελτίωση των εργασιών των δύο κατηγοριών δομών. Δεύτερον, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την υφιστάμενη σύνδεση τη ημερήσια διάταξη ολομέλεια στο Στρασβούργο και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η δράση αυτή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιλάβει την άσκηση περισσότερου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή του Συμβουλίου των Υπουργών, συγγνώμη, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κατά κάποιο τρόπο ως πρόδρομοι κριτές. Οι συζητήσεις των Πρωθυπουργών με τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν να περιλάβουν και τις ημερήσεις διατάξεις ε, του Στρασβούργου και των Βρυξελών. Αν εκμεταλλευτούμε τις τεχνικές δυνατότητες της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε την ε, απομάκρυνση της κοινή γνώμης από τις δραστηριότητε μας και τη μείωση του ενδιαφέροντος για μας. Και σας μιλώ ως βουλευτής από την περιφέρεια που θα ήθελε να μπορεί να συναντηθεί με την Επιτροπή ε, ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια θέση του Κοινοβουλίου μας και όχι στην Λισαβόνα. diskutiert worden. Κοιτάξτε, παράλληλε συζητήσει έγιναν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά ε, Κοινοβούλια. Τώρα, κατά πόσο αυτέ γίνεται στο Συμβούλιο, το αμφισβητώ. Τέλο πάντων, κύριο Άλιστα. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει ένα βαθμό ε, υποκρισία στην έκθεση αυτή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Επιτροπή μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να υπονομεύσουν τελικά τα εθνικά κοινοβούλια όσο δυνατόν, περισσότερο. Και μάλιστα προσπαθούν να πάρουν αρμοδιότητες από τα κοινοβούλια αυτά και να φέρουν τι αρμοδιότητες αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και Τώρα ξαφνικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ πιστεύουν ότι έχουν νικήσει τη μάχη, λένε ότι θα πρέπει να δείξουμε και μια κάποια μεγαλοψυχία. Ουσιαστικά αυτό προσπαθεί να κάνει η έκθεση αυτή. Είναι σαν να λέμε πια στο, στα εθνικά κοινοβούλια, κοιτάξτε, έχετε πια μια επιλογή μπροστά σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην κίτρινη ή την πορτοκαλή κάρτα, ενώ στην πραγματικότητα τους δείχνουμε μια κόκκινη κάρτα. Ας έρθουμε λέμε ότι θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους, ότι θα τους συναντούμε όλο και περισσότερο. Στην πραγματικότητα έχουμε κλέψει τις αρμοδιότητές τους. Λέμε τώρα ότι θα είμαστε καλοί μαζί τους. Νομίζω ότι αυτή η νοτροπία τελικά κρύβεται πίσω από την έκθεση αυτή και νομίζω ότι αν διαβάσει κανείς αντικειμενικά την έκθεση αυτή θα καταλάβει τι κρύβεται πίσω από την έκθεση. Και πιστεύω ότι είναι αρκετά υποκριτική η στάση η οποία διατηρείται στην ε, έκθεση αυτή μέσα στα άρθρα τη έκθεση αυτή. Ενώ στην πραγματικότητα, το πανλαμβάνω, θεωρώ ότι έχουμε πάρει αρμοδιότητε από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να τι φέρουμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Ενρίκε. Στο κυρίου Άλιστερ, βέβαια, αυτή. Ενρίκε. Ε, Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, μια και είναι η πρώτη φορά που μιλώ στην αίθουσα που έχει το όνομα του Γιώζεφ Αντάλ, αυτής τη μεγάλης προσωπικότητας, δημοκράτη, ευρωπαϊστή Ούγγρου, που τον είχα γνωρίσει την εποχή της μεταπολίτευσης στην Ουγγαρία, έναν ανθρώπου που τιμά την Ευρώπη, να το αναφέρω αυτό. Μία σχεδόν προϊστορικού χαρακτήρα παρατήρηση, που έχει σημασία όμως ως προηγούμενο και δεν το αναφέρει η έκθεση Μπροκ. Το εξής. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν έπαιζαν άμυνα μόνο εναντί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνέβαλαν με πολύ σημαντικό τρόπο και στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Σας θυμίζω ότι το 1990 επί προεδρίας μου συναντήθηκε στο Μοντετσιτόριο της Ρώμης μια διάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών της κοινότητας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι γνωστές ασύζ της Ρώμης καθοριστικού χαρακτήρα για την προπαρασκευή της συνθήκης του Μάστρεχτ. Στη διάσκεψη αυτή ο εισηγητής εξ του όλων των κοινοβουλίων ήταν ο πρόεδρος της Βουλής του Βελγίου το αίτημα που υποβάλαμε δε όλα τα κοινοβούλια να και που επέτρεψε να προχωρήσουμε στη συνθήκη του Μάστεχτ ήταν ομόφωνο. Δεν παίζουμε λοιπόν η μεν έναντι των δε, τον δε το εθνικ, τα εθνικά κοινοβούλια έναντι του Ευρωπαϊκού. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό να το θυμίσουμε αυτό το γεγονός που είχε σημαντικό ιστορικό χαρακτήρα. Μετά, στο σημείο 1 που μιλάει για το δικαίωμα συμμετοχής να σας πω ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με ένα σανσέρ, η αρχή της επικουρικότητας δεν κατεβαίνει μόνο, αλλά πρέπει να και να ανέβει. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε την διενεργή αυτή διάσταση σε μια έκθεση. Δεν Ξέρω αν υπάρχει χώρος. Πιστεύω ωστόσο ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι μαζί δουλεύουμε. Όχι ο ένας κοντά στον άλλον. Ευχαριστώ. ο Αντρέ Σεβερίν. 7 έχουμε. Και μετά θα κλείσω την ε, συζητηση τρια Τρία-τέσσερα λεπτά παρακαλώ να τελειώνετε. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούριο σίγουρα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια της ε, Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ε, Ορισμένες από τις ιδέες λοιπόν είναι ειδικά, ιδιαίτερα ξεκάθαρες, ιδιαίτερα σαφείς, δεν υπάρχει κάτι φοβερό το οποίο πρέπει να προσθεθεί στην έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι γενικά καλή, αναφέρεται σε διάφορες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί καλύτερα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα ήταν σωστό για μας κάπου να λέμε με πιο σαφή τρόπο ποιος είναι ο στόχος του όλου χειρήματος. Ακριβώς για να αποφύγουμε τους ε, φόβους αυτούς ή τις ε, επικρίσεις αυτές που εξέφρασε ο κύριος Άλιστερ πριν από λίγο, σχετικά δηλαδή με την ε, υποκρισία, με την υποκριτική μας δίθεν στάση. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα σε κάποιο σημείο ότι κανείς δεν έκλεψε τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων. Αποφασίσαμε ουσιαστικά να εξασκήσουμε μαζί τις κυρίαρχες αυτές αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ληφθεί κατά τρόπο επίσημο και αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να μοιραζόμαστε καθήκοντα όσον αφορά τον νομοθετήν και όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την παρακολούθηση προκειμένου να καταφέρουμε δηλαδή να μοιράσουμε, να κατανείμουμε καλύτερα τη δουλειά μας, αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να βρούμε κάποιους τρόπους συνεργασίας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει κάπου να λέγεται ξεκάθαρα στο κείμενο, ποιος είναι ο στόχος του όλου εγχειρήματος. Και κάτι ακόμα, στόχος επίσης του εγχειρήματο, είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες των εθνικών κοινοβουλίων όταν εμείς νομοθετούμε και τα εθνικά κοινοβούλια με τη σειρά τους να καταλάβουν καλύτερα τι κάνουμε εμείς εδώ όταν εμείς εδώ νομοθετούμε. Κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μία επικοινωνία που θα οδεύει προς τη σύγκληση και όχι προς την απόκληση και να φέρουμε στην επικοινωνία με τους ψηφοφόρους μας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνεται μια σωστή διάκριση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων και χωρίς να αλλάξουμε πάρα πολύ το κείμενο, θα πρέπει σε κάποια σημεία να φαίνεται ξεκάθαρα ποιο είναι ο στόχο του ελεγχειρήματος, ποιο είναι ο στόχο τη έκθεση αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να διασκεδάσουμε οποιασδήποτε ανησυχίε, αμφιβολίες και σε καμία περίπτωση θα μπορεί κανεί να διατείνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκλεψε εθνικέ αρμοδιότητες, αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, όταν σπούδαζα νομική, έμαθα τότε ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Αυτή η σχέση είναι αυτόματη. Από τη στιγμή που έχει κανείς ένα δικαίωμα, έχει και μία υποχρέωση. Και στην έκθεση αυτή δεν γίνεται καμία αναφορά στις υποχρεώσεις οι υποχρεώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιωμάτων, συνδέονται άμεσα με τα δικαιώματα αυτών, αυτού του Κοινοβουλίου. Αναφερόμαστε μόνο σε δικαιώματα χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε υποχρεώσεις. Μία υποχρέωσή μας θα ήταν να εξασφαλίσουμε την ε, συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κατά το δυνατό βέβαια, όσο αυτό είναι δυνατό, είδαμε ότι σε ορισμένε χώρε τα εθνικά κοινοβούλια νομοθετούν χωρί να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τις βασικές νομοθετικές στάσεις που εκφράζονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ψηφίζονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συναντάμε πάρα πολλές περιπτώσεις πάρα πολλά προβλήματα όταν προσπαθούμε στη συνέχεια στις χώρες αυτές να μεταφέρουμε και να εφαρμόσουμε την κοινοτική νομοθεσία. Ένα μόνο παράδειγμα είναι αυτό για να σας τονίσω ότι σε καμία περίπτωση ούτε τα εθνικά δηλαδή κοινοβούλια μπορούν να έχουν δικαιώματα χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες ανάλογες υποχρεώσεις. Μολονότι μπορεί να μην γίνεται σαφή αναφορά στι υποχρεώσει αυτέ στη συνθήκη, αυτέ υπάρχουν από τη στιγμή που θεσπίζονται δικαιώματα. Και κάτι ε, τελευταίο θα ήθελα να πω. Να πούμε καταρχάς πρώτον ποιος είναι ο στόχος του εγχειρήματο αυτού, επαναλαμβάνω για να αποφύγουμε παρανοήσεις και για να δώσουμε μια καλύτερη προοπτική τόσο για τα εθνικά κοινοβούλια όσο και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια για τη μελλοντική μας συνεργασία. Πρώτον αυτόν λοιπόν και δεύτερον να καταφέρουμε να αναφερθούμε σε κατα, κατά κάποιο τρόπο στην συμπεριφορά που περιμένουμε από τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν έχουν μόνο αυτά δικαιώματα στη συνεργασία μαζί μας, αλλά και εμείς έχουμε δικαιώματα όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την έκθεση αυτή, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ καλή. Δεν είμαι σίγουρος ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να μιλήσει για υποχρεώσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά μάλλον για δυνατότητες συνεργασίας και νομίζω ότι το σημείο 8 περιλαμβάνει κάποια παραδείγματα για τα οποία, με τα οποία μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία αυτή. Κύριε Μότ. Ah, Ξέρετε, δεν είμαι συνηθισμένο στις νέες τεχνολογίες. Συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή, πρόεδρε. Κάτι λείπει στην έκθεση. Διαφωνώ όμως ουσιαστικά για το τι λείπει. Όπως το διαβάζω, το κείμενο δεν έχει τίποτα για το γεγονός ότι η Ένωση αναγνωρίζει την πλήρη κυριαρχία των κρατών μελών. Ούτε καν στις καθημερινές σχέσεις μεταξύ Ένωσης κρατών μελών. Έγιναν δύο επισκέψεις μελών του Κοινοβουλίου στην Πράγα τις τελευταίες εβδομάδες. Και στις δύο καταφέραμε να αφήσουμε μέλη του Κοινοβουλίου να συμπεριφερθούν με τρόπο που μόνο προσβλητικό και υπεροπτικό προς ένα κράτος μέλος θα χαρακτηρίζα. Προσπάθησαν να πούν και να απειλήσουν την τσεχική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξαγάγει την προεδρία της. Το ίδιο επαναλήφθηκε και στην πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια μετά την έναρξη της τσεχικής προεδρίας. Ε, αξιο... Απαράδεκτο είναι το να θεωρείτε ότι το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα στη συμπεριφορά κυρίαρχων κρατών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταφ. Γεια σας. Εγώ μιλάω από την ομάδα των Βρετανών, εκεί τη γωνίτσα πίσω. Αυτά που θα πω όμως απέχουν κάπως από αυτά που, που είπαν οι συμπολίτε μου που μίλησαν νωρίτερα. Κάποιοι από εμά περάσαμε πολύ χρόνο και προσπάθειες για να προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να τα ενημερώσουμε για το πώς πάνε τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι βέβαια λογικό να υπάρχει μια κάποια ένταση μεταξύ του κεντρικού, του ομοσπονδιακού και των ομόσπονδων κοινοβουλίων. Αλλά η ένταση αυτή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φαίνεται και να είναι δημιουργική, να λειτουργεί με οργανωμένο τρόπο, χωρίς να προκαλεί συγκρούσεις. Και πρέπει να σας πω ότι οι διαδικασίες που σταδιακά τέθηκαν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αρχίζουν και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτό σίγουρα συμβαίνει με την Κόζακ που έγινε ένα φόρουμ με πολύ περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο από ό,τι πριν. και νομίζω ότι η έκθεση Μπροκ ε, καταφέρνει να το περάσει αυτό το νόημα. Στην παράγραφο 2, Πρόεδρε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μνήμα σε αυτό το αναεξάμεινο φόρουμ που δημιουργήθηκε για να παρακολουθήσει τις, τις συνταγματικές διαπραγματεύσεις. Πάντα θα μπορούσαμε να προωθήσουμε το ενδεχόμενο ειδικών συναντήσεων μεταξύ πολιτικών ομάδων και στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το να προσπαθήσουμε όμως να το οργανώσουμε χωρίς ε, δηλαδή πιέζουμε την ημερήσια διάλεξη χωρίς να έχουμε πραγματικά πολιτικά θέματα να συζητήσουμε αναπερίπτωση. Εφόσον δεν υπάρχει περί, κάποια διακυβερνητική ή νομίζω ότι εκτός διακυβερνητικής, περίοδου διακυβερνητικών, πιο ενδεδειγμένο θα ήταν να, να παραμένουμε στην συνεργασία των ε, καθήλυνα αρμοδίων επιτροπών. Επιπλέον, η Επιτροπή Εξωτερικών θα μας στείλει μια εξαιρετική έκθεση σχετικά που θα εξετάσουμε ε, εν ευθέτω χρόνο. Την περιμένουμε. Πάντως, το φόρουμ, το, το κοινοβουλευτικό φόρουμ ξεκίνησε με την περίοδο περισυλλογής. Αλλά θέσατε μια σειρά, θέτηκα μια σειρά μεγάλων θεμάτων, αλλαγή κλίματος, στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Κύριος Μποτόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Μια γενική παρατήρηση και τρεις ερωτήσεις προς τον κύριο Μπρόκα. Η γενική παρατήρηση έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι από νομικής πλευρά συμφωνούμε όλοι ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έχουν χάσει αρμοδιότητες. Ουσιαστικά χάσανε, αν θέλετε, αρμοδιότητες εκεί που είχαν αποκλειστική αρμοδιότητα. Άλλο όμως αυτό Άλλο το να έχουμε κοινέ πλέον αρμοδιότητε ή να μοιραζόμαστε αρμοδιότητε και άλλο να λέμε ότι εθνικά κοινοβούλια έχουν χάσει αρμοδιότητε. Και όσον αφορά στη συνέχεια τη συνεργασία για τα, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Στην παράγραφο τώρα 6. Ο κύριος ε, Μπρόκ αναφέρεται στους επικεφαλείς εξειδικευμένων επιτροπών. Γιατί όμως μόνο στα δύο αυτά ε, θέματα, πολιτικές ελευθερίες και εξωτερικές υποθέσεις, για ποιο λόγο να μην συμπεριλάβουμε και τα συνταγματικά θέματα, εφόσον είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιο λόγο να μην έχουμε και άλλες επιτροπές σε αυτή την παράγραφο αυτή. Στη συνέχεια για την παράγραφο 8 για το ζήτημα των υποχρεώσεων, στο οποίο αναφέρθηκε και άλλος συνάδελφος, να θέσουμε τις υποχρεώσεις, να αποσαφηνίσουμε τις υποχρεώσεις των εθνικών κοινοβουλίων. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αμφιβάλλον μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει στα εθνικά κοινοβούλια έχετε περισσότερες υποχρεώσεις. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι, κοιτάξτε, να τι γίνεται σε κάποια εθνικά κοινοβούλια. Ενδεχομένως και εσείς χι εθνικό κοινοβούλιο να αναλάβετε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ενδεχομένως να καλέσετε ε, και εσείς με τη σειρά σας, όπως κάνουν άλλα κοινοβούλια, ε, βουλευτές από άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια στην παράγραφο 19 συστηματική παρακολούθηση του προνομοθετικού διαλόγου. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα, λίγο πιο ουσιαστικά. Νομίζω ότι να γίνεται απλώς μία αναφορά στην συστηματικότερη αυτή παρακολούθηση του διαλόγου είναι κάτι το αρκετά αόριστο. Ίσως θα έπρεπε εδώ να βάλουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε αυτή η παρακολούθηση να γίνει πιο συστηματική. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κόρμπετ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στις Επιτρέψτε μου να το πω αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Άλιστερ. Δεν νομίζω ότι έπεισε κανέναν εδώ. Δεν ξέρω ε, τι τον όθησε να πει αυτά που είπε ίσως το ίντερνετ, το web streaming το, και οι κάμερες δεν βλέπω να έμεινε εδώ, να κάθισε εδώ, να, ακού, να ακούσει και καμιά άλλη άποψη ε, διαφορετική από τη δική του. Σε λιγότερο από μισή ώρα εξεφανίστηκε, Αλλά να καλό παράδειγμα των ε, Βρετανών ευρωσκεπτικιστών είναι ο κύριος αυτός όταν είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την άποψή του κλέβει, προσπαθεί να κλέψει αρμοδιότητες από τα εθνικά κοινοβούλια ε, ε, αυτό προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα εμείς εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αρμοδιότητες ε, τέτοιες που αποφάσει που τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια μας ανέθεσαν όταν ε, κύρωσαν τις ε, συνθήκες υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα μοιράζονται τα εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια συμφώνησαν για τις εξουσίες ή τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και εμείς υποστηρίζουμε τις προσπάθειές του τους να ενημερώνονται καλύτερα κτλ. κτλ για να μπορούν να με παρακολουθούν τους υπουργούς τους τι κάνουν στην Ευρώπη και τα Λοιπόν αυτές ε, οι, οι αρμοδιότητες αν θέλετε και οι εξουσίες των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι συμπληρωματικές δεν είναι αντιπαρατίθενται οι μεν στις δε από εκεί και πέρα το να παρουσιάζονται τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσίασε ο κύριος Άλιστερ είναι τουλάχιστον διεστρέβλωση της πραγματικότητας έτσι δεν το συζητάμε θα ήθελα αυτό να περάσει τα πρακτικά ε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος για όλους αυτούς και εκ μέρους όλων αυτών που παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να τονιστεί ότι δεν κλέβει αρμοδιότητες Εθνικών Κοινοβουλίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ε, απλώς ε, ε, βοηθάει στην παρακολούθηση και την, ε, τον έλεγχο των, της εκτελεστικής εξουσίας αν θέλετε γιατί δεν είναι πια μόνοι τους αυτοί όσον αφορά το νομοθετικό έργο που εκτελούν και τα λοιπά ο επόμενος ομιλητής Μίλησε ο κύριος ε, Μπαρόν Κρέσπο για τον Γιώζε Φάνταλ θα ήθελα κι εγώ λοιπόν να σας καλέσω την άλλη πέμπτη πρωί σε μια ε, σε μια συνάντηση, αναμνηστική συνάντηση, ε, σε μια συνάντηση στο, ακριβώς για τον κύριο Άνταλ ο Ιωζεφ Άνταλ έκανε δύο σημαντικά πράγματα ξεκίνησε την διάλυση του Συμφώνου της Βασοβίας και ξεκίνησε την Συμφωνία Βίσεχαρτ που ήταν η πρώτη συμφωνία των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης για ενόψη της μελλοντικής ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτησα να μιλήσω για ένα θέμα στην έκθεση Μπροκ που αναφέρεται στο σημείο 8 όπου καλωσορίζουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που επιτρέπουν σε μέλη του Κοινοβουλίου να έχουν περισσότερα δικαιώματα στους εθνικούς νομοθέτες. Αυτό το κείμενο θεωρητικά παρουσιάζεται, αλλά εγώ μπορώ να σας θυμίσω το, την πρακτική στο Ουγγρικό Κοινοβουλίο και ίσως επειδή είμαστε καινούργοι έχουμε και κάποια πλονεκτήματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα που αναφέρετε τα έχουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Μπορούμε να κληθούμε και να μιλήσουμε για οποιοδήποτε ζήτημα στο Εθνικό Κοινοβούλιο που αφορά ευρωπαϊκά θέματα. Δηλαδή, το, εθνικό, το, εθνικό, μας κοινοβούλιο έχει κατάλογο των κειμένων που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, τα καταγράφει αυτά και, στην ομολο... και μπορούμε να μιλήσουμε στην Ολομέλεια για τα θέματα αυτά. Επίση, μπορούμε να μιλήσουμε, να παραστούμε και να μιλήσουμε σε όλε τι επιτροπέ, ιδιαίτερα δε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα έλεγα λοιπόν να ενισχύσουμε το κείμενο λέγοντα ότι Υπάρχουν ήδη παραδείγματα τέτοιων πρακτικών σε άλλα εθνικά κοινοβούλια, δίνοντας και κάποια παραδείγματα. Γιατί ξέρετε τώρα αρχίζει το ανάποδο να πάρουν πίσω τα δικαιώματα. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα παραδείγματα αυτά και για άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Πριν τον Έλμαρ Μπρόκ, να καλωσορίσω τον κύριο Γιούρη. από την Σλοβενία, πρώην Πρωθυπουργό. Καλώς ήλθατε. Νόμιζα ότι ήσασταν από την Επιτροπή Γιούρη, την νομική, αλλά έτσι σας λένε το επίθετό της. Το επίθετό σας. Έλμαρ, άκουσες πολλά πράγματα, ξέρεις και τι υπόθηκε όταν ήσουν έξω. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που έκαναν ε, παρεμβάσεις και θα ήθελα να αναφερθώ, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Νταφ ε, και θα ήθελα να του πω ότι δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με τους ε, Βρετανούς δεν με ενοχλούν ιδιαίτερως ακόμη και αν εκφράζουν απόψεις ε, οι οποίες ε, μου είναι μάλλον ξένες. Εν πάση περιπτώσει η συνθήκη της Λισαβόνας κυρίες και κύριοι είναι ουσιαστικά η συνθήκη του Κοινοβουλίου έτσι και νομίζω ότι αυτό όταν λέω το κοινοβούλιο είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια που περιλαμβάνονται εδώ όταν ο συνάδελφος Σεβερίν ε, θέτει το θέμα των υποχρώσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων όντως ε, πρέπει να του απαντήσω ότι η συνθήκη αφήνει κάποια παράθυρα ανοιχτά από την άλλη μεριά όμως εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στα Εθνικά Κοινοβούλια ε, υπάρχουν όντως δυνατότητες όπως ελέγχθη όχι υποχρεώσει δυνατότητες ε, και αυξήθηκαν αυτές πάρα πολύ με την συνθήκη της αυξάνονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας και επίσης η έγκαιρη ενημέρωση που προβλέπεται το να μπορεί κανείς να γνωρίζει έγκαιρα ορισμένα πράγματα ε, πότε αρχί, όταν αρχίζει η νομοθετική δουλειά δηλαδή στο Συμβούλιο να μαθαίνουν οι επιτροπές περί τίνος πρόκειται αυτή η έγκαιρη ενημέρωση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική είναι ε, κάτι ε, που βεβαίως μπορούν να το αποφασίσουν mm. όχι μπορούν να τα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω σε αυτό Στο, στη Γερμανία λόγου χάρη ε, το άρθρο 23 του συντάγματος επιβάλλει κάτι τέτοιο απ' την άλλη μεριά άμα κοιτάξετε την έκθεση του Ιρλανδικού της Ιρλανδικής Βουλής του Νοεμβρίου ε, που αναφέρεται στο δημοκρατικό έλλειμμα και τους τρόπους καταπολέμησης της κατάστασης αυτής και Αναφέρεται η έκθεση αυτή σε ανάγκη, ανάγκη στην αναγκαιότητα στενότερων σχέσεων και συντονισμού με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, φαντάζομαι ότι αυτά που λένε οι Ιρλανδοί ισχύουν και, και για όλους τους άλλους. Όντως ε, ε, νομίζω ότι σε πάρα πολλά κράτη-μέλη η Βουλή ακολουθεί την σωστή το σωστό δρόμο αν θέλετε σχέσεις με το κοινοβούλιο τώρα βίντεο conference αναφέρθηκε εδώ μιλάμε για την, ε, πριν από την έκδοση νομοθεσίας κτλ κοιτάξτε ε, ε, από εκεί και πέρα η τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης είναι άλλο πράγμα. Ορισμός της ημερήσιας διάταξης, η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ε, είναι τεράστιο δικαίωμα, πολύ σημαντικό δικαίωμα αν θέλετε του, της Βουλής. Υπάρχουν ε, ε σε ορισμένες χώρες ε, κοινοβουλία τα οποία δεν είναι μόνα αυτά υπεύθυνα για τον κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης. Ε, αυτό είναι τεράστια απώλεια αν θέλετε δικαιώματος. Λοιπόν το λέω αυτό γιατί δεν είναι αστείο το ποιος ορίζει όχι την ημερήσια διάταξη. Τώρα, ο κύριος Μόουτ τι μου είπε, μου είπε ότι δεν αναφέρεται εδώ η εθνική κυριαρχία και αυτονομία των κρατών μελών. Συγγνώμη, η συνθήκη της νίκαιας δίνει στα εθνικά κοινοβούλια πολύ λιγότερες δυνατότητες και δικαιώματα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυξάνονται σημαντικά τα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων. Από εκεί και πέρα η εθνική κυριαρχία δεν νομίζω ότι αμφισβητείται και, και δεν νομίζω ότι ε, χρειάζεται να πούμε τίποτα για την εθνική κυριαρχία αν δεν θέλουμε να γίνουμε γελοί σε τελευταία ανάλυση. Στο συνάδελφο, θα ήθελα να παρακαλέσω τον συνάδελφο Μποτόπουλο να με βοηθήσει για ο κύριος Μπουτόπουλος λοιπόν να με βοηθήσει εδώ στην παράγραφο 19 για τη συστηματικότερη παρακολούθηση του διαλόγου. Τον παρακαλώ ε, να μου κάνει κάποια πρόταση σχετικά και για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα να πω μερικά πράγματα για τις συναντήσεις τις διακοινοβουλευτικές. Κοιτάξτε, εγώ δεν αμφισβητώ ότι κάποιες συναντήσεις αυτά το interparliamentary φόρα και τα λοιπά είναι σημαντικά βήματα ανταλλαγής απόψεων. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να ε, γίνω, οργανώνονται αυτού του είδους οι συναντήσεις αλλά εκτάκτος, ad hoc άμα υπάρχει ανάγκη αλλά το να συστηματικοποιηθούν, να θεσμοθετηθούν και αυτή είναι η γαλλική ιδέα μετά τη συνέλευση της, ε, των συναντήσεων αυτών ε, αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό το να είναι μόνο μόνιμες ε, θεσμοποιημένες και μόνιμες οι συναντήσεις αυτές ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται δεν, είναι, δεν βελτιώνει και πολύ τα πράγματα ε, γι' αυτό δεν μπήκε στο σημείο 2 όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ε, οι ε, τεχνικές επιτροπές συναντιούνται πολύ συχνά και τα προβλήματα επιλύονται με αυτόν τον τρόπο τώρα για κάποιους να πω μερικά πράγματα για τη μεταρρύθμιση του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον ε. Ε, γιατί αναφέρθηκε και αυτό εγώ νομίζω ότι η ευθύνη ε, για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και στο μέλλον είναι ε, ευθύνη των επιτροπών, της επιτροπής, των προέδρων των επιτροπών αλλά δεν πάω παραπέρα, δεν μιλώ για συνδιάσκεψη των προέδρων και τα λοιπά. Όχι, εγώ νομίζω ότι ε, η, η διάσκεψη των προέδρων ουσιαστικά ε, ε, θα πρέπει απλώς να μαθαίνει τι αποφάσισαν οι πρόεδροι οι, των επιτροπών ή η διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε δηλαδή μεγαλύτερο μεγαλύτερο βαρύτητα σε ορισμένα πράγματα από αυτοί που έχουν ε, και να μην κάνουμε μονιμότερα κάποια βήματα τα οποία δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνιμα. Νομίζω ότι οι επιτροπές στην οποία λαμβάνουν μέρος τα, οι βουλευτές ε, και αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι είναι το κύριο όργανο αν θέλετε του Κοινοβουλίου. Ε, Εν πάση περιπτώσει ε, αυτά κύριε Πρόεδρε δεν θα πω παραπάνω καταθέστε τις τροπολογίες σας για να φτιάξουμε σύντομα και το οριστικό κείμενο για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ λέει ο Πρόεδρος. Η έκθεσή σας είναι όντως πολύ σημαντική ε, η σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια είναι πραγματικά ε, πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, η κατάθεση τροπολογιών μέχρι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται στις 4 Μαρτίου 12 η ώρα του μεσημέρι και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Προχωρούμε στο επόμενο ε, θέμα της ημερήσιας διάταξης την, ε, για την ε, πώς τη... ομάδα προβληματισμού της οποίας προεδρεύει ο Φελίπε Γκοντζάλες ε, θα δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της ομάδας αυτό, αυτής προβληματισμού με τιτλο οριτζοντε Οριτσόντε 2020-2030 ε, νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεων μέσα στην ομάδα αλλά και η δική μας ενημέρωση σχετικά είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας γιατί πραγματικά φαντάζομαι ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πάρα πολύ ε, σοβαρές. Ο κύριο Βέστενμπορκ, ο Κάρλος και τον χαιρετίζω βρίσκεται ήταν, είναι παλιός συνάδελφος και χαίρομαι ιδιαίτερα τη συμμετοχή του. Ε, είναι πάρα πολύ καλό το ότι είμαστε όλοι μαζί σήμερα. Δεν θέλω να καθυστερήσω. Χαιρετίζω απλώς το γεγονός ότι η Ευρώπη ε, δεν δουλεύει μονάχα με την καθημερινότητα αλλά και με το μέλλον προσπαθεί να φανταστεί το μέλλον ε, μέχρι τώρα μας λέγανε οι Αμερικανικοί ότι οι πρόεδροι οι Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι βλέπανε το μέλλον και είχαν οράματα για τη χώρα τους και τα λοιπά ε, και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φτιάξει ούτε μια καινούργια συνθήκη παραμένει στα παλιά και δεν ξέρω ότι όχι, εγώ νομίζω ότι η ομάδα προβληματισμού από την προεδρία του κ. Κοντζάλε κάνει σοβαρότατη δουλειά και πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον συζητήσα και αυτές που θα γίνουν εδώ να γίνουν και με τους Ευρωπαίους πολίτες με την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλά, μα, πολλές, μα πολλές προσδοκίες. Φελίπε Γκονζάλες έχει το λόγο. Ε, amigos parlamentarios. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το να διευνήσει κανείς το μέλλον με το βαθμό της αβεβαιότητας στον οποίο ζούμε μπορεί να είναι τόσο δύσκολο που να οδηγεί σε μελαγχολικές με συμπεριφορές. Το να λέμε για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη του 2020 είναι εξίσου δύσκολο με το να μιλά κανείς για το παρελθόν στην Ισπανία. Είναι εξίσου απρόβλεπτο όπως και το παρελθόν μας. Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω, αυτό είναι βασική προφύλαξη ότι χτες είχαμε την πρώτη συνάντηση συζήτηση της ομάδας προβληματισμού. Μια συζήτηση που, που έκανε κατά βάση background και ανάλυση του γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση, αυτό που λέω για το περιεχόμενο στην, στις συζητήσεις που έχουμε είναι προσωπικές απόψεις, όχι απόψεις της ομάδας προβληματισμού. Δεν θέλω να δεσμεύσω την ομάδα των 12 μελών με κάτι που ακόμα δεν ξεκινήσαμε καν να διακρίνουμε και να δουλεύουμε. Προχωρήσαμε μεθοδολογικά στη μέθοδο εργασίας και κάποιες, σε κάποιες από τις προτεραιότητες, προτεραιότητες και το περιεχόμενο και χθε είχαμε τις πρώτες συζητήσεις στην ομάδα για την παρούσα κατάσταση και τα στοιχεία από τα οποία θα μπορούσε, στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί ο προβληματισμό για το μέλλον. Αυτό θέλω να, αυτό θέλω να πω ότι η ομάδα έχει τη βούληση να προβεί σε μια ανάλυση στρατηγικών στόχων εν ώψη του ορίζοντα 2020 που θα είναι μια ενεργή ενεργητική στρατηγική που δεν θα λειτουργεί αμυντικά. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να διαμορφώσουμε το μέλλον απαντώντας ή για να βοηθήσουμε τέλο πάντων να διαμορφώσουμε το μέλλον υπό τις αιρέσεις βέβαια της προβλεψιμότητας απαντώντας σε δύο μεγάλα θέματα. Ένα, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει σπουδαιότητα για τον πολίτη της ή προς τα αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σημασία, σχετική σημασία για τον πολίτη και πώς να κερδίσει σημασία έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Πώς σχετίζεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινήσαμε βάσει ενός ψηφίσματος του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πριν από 14 μήνες στη Λισαβόνα. Ε, της Λισαβόνα, η... αυτό έγινε την επαύριο της υπογραφής της συνθήκης της Λισαβόνας στις Βρυξέλλες. Πάντως εκείνη τη στιγμή η υπογραφή της συνθήκης ε, επέτρεψε στο Συμβούλιο να σκεφτεί ότι είχαν λυθεί τα θεσμικά ζητήματα με το βαθμό ικανοποίησης του καθενός από το περιεχόμενο της συνθήκης. Είχαν λυθεί ωστόσο τα θεσμικά εργαλειακά αν θέματα λειτουργίας της Ευρώπης με την σημερινή μορφή της. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε μέχρι την εκλογή, την επιλογή των 12 μελών της ομάδας, μην ξεχνάτε ότι στην πρώτη φάση επέλεγησαν τρία άτομα, πρόεδρος και δύο αντιπρόεδροι, και μετά οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί Γαλλικής Προεδρίας. Ένας χρόνος λοιπόν πέρασε τι θέλω λοιπόν να πω για να εισαγάγω τη συζήτηση στο υφιστάμενο πλαίσιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που έγινε από τη στιγμή που λήφθηκε η απόφαση δημιουργίας μιας ομάδας προβληματισμού με έναν ε, στρατηγικό ορίζοντα 2020-2030, εγώ θεωρώ πιο φρόνιμο να μιλήσουμε για το 2020, γιατί οι μόνοι που μιλάνε συνεχώς για το 2020 30 είναι οι Κινέζοι. Οι Ευρωπαίοι μιλούν πιο βραχυπρόθεσμα για να δημιουργήσουν ε, ε, ανέκδοτα. Ε, αυτό που βλέπουμε λοιπόν ε, με σε αυτό το εν του χρονικού αυτού οριζοντά από την λήψη απόφασης μέχρι τώρα βρισκόμαστε στα πλαίσια μιας θεσμικής κρίσης που προέκυψε από την απόρριψη της συνθήκης της Λισαβόνας από την Ιρλανδία. Δεν κρίνω την απόφαση, αλλά σας λέω ότι έχουμε μια θεσμική κρίση. Ταυτόχρονα κάλπαζε η οικονομική κρίση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε επίγνωση ακόμα ότι αυτή η, οικονομική, ότι η κρίση που είχε ξεκινήσει από τα subprime τον είπα ότι θα επηρέαζε και την Ευρώπη. Το Νοέμβριο του 2007 μάλιστα πιστεύαμε ότι το πρόβλημα των subprimes ήταν ένα, ευρωπαϊκό, ένα αμερικανικό, συγγνώμη, όχι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν το πίστευαν όλοι αυτό, αλλά εν γέννη οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες πίστευαν ότι η κρίση δεν θα επηρέαζε ή την Ευρώπη ή δεν θα την επηρέαζε τέλος πάντων με τόσο βαθύ τρόπο όπως την επηρέασε. Τότε λοιπόν δεν θεωρούσαμε δεν θεωρήτο. Και τότε και μήνες μετά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού που πέρασε, δεν εθεωρείτο ότι η κρίση του οικονομικού συστήματος ήταν συστημική. Όλοι νόμιζαν ότι ήταν αμερικανική. Οι συστημικές κρίσεις είναι μάλιστα μία από τις πιο παράδοξες συστημικές κρίσεις. Είναι κρίση του συστήματος αλλά δεν υπάρχει εναλλακτικό σύστημα υποκατάστασης. Δεύτερο θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτον, θεσμική κρίση. Δεύτερον, οικονομική κρίση. Οι συνέπειες της οποίας στην πραγματική οικονομία είναι σκληρές, σκληρότατες, καταστρεπτικές θα έλεγα. Χάσαμε 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Είναι συστημική και άρα επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Διαδοχικά, διάφορες περιοχές του κόσμου άρχισαν να αποδέχονται ότι η κρίση τι αφορά. Η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική, η Ασία. Η κρίση λοιπόν είναι κρίση του συστήματος. Τρίτο θέμα. Πέραν της θεσμικής και της οικονομικής κρίσης, με πολύ σκληρές συνέπειες για την παραγωγική ή πραγματική όπως τη λέμε οικονομία, που οδηγεί σε μια παγκόσμια ύφεση, για να μην σας πω σκληρή ύφεση, που απαιτεί συντονισμένη δράση. Τρίτο στοιχείο. Όσο εξελίσσεται και οριζόταν η εντολή της ομάδας, με μια, με μια σαφή αναφορά του η εντολή μας διαμορφωνόταν με μια σαφές, περιεχόμενο του ότι δεν πρέπει να αθήξουμε αλλά σαφέ περιεχόμενο του τι πρέπει να εξετάσουμε. Μας λέγανε, μη μιλάτε για τα θεσμικά γιατί τα έλυσε η Λισαβόνα, μη μιλάτε για τα οικονομικά γιατί αυτά είναι δική μας αρμοδιότητα, πού να πάμε. Αυτή ήταν η εντολή που είχαμε. Πριν ξεκινήσει η δουλειά της ομάδας προβληματισμού, που όπως είπα τώρα μόλις πρώτο συναντήθηκε, γιατί δεν είχε ούτε καν προϋπολογισμό για να συναντιόμαστε πριν τη συνάντηση έρχεται η θεσμική κρίση, η συστημική κρίση στην οικονομία και μια κρίση στην ασφάλεια, διότι στην, ε, στην εντολή μιλάει, η εντολή μιλάει για τις απειλές στην ασφάλεια της Ευρώπης, μιλώντας για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Σωστό, αρκετά σωστό. Πρόκειται για τις πιο μόνιμες, ορατές απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά καθοδόν εκ νέου εμφανίστηκε μια κρίση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας που σχετίζεται κάπως και με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αργότερα, τις τελευταίες εβδομάδες, είχαμε μια κρίση στην Εγγύς Ανατολή, Μέση Ανατολή τέλο πάντων, για την Αμερικανική οπτική γωνία, μιας ενός τέτοιου μεγέθους και οξύτητας που ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συνέπειες θα είχε. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία συνέπεια σίγουρη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να πληρώνει τα έξοδα της ενοικοδόμησης, πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Γάζα. Επιπρόσθετο στοιχείο που ήρθε και έκατσε από πάνω. Έχουμε δύο ζητήματα που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως προβλήματα που περιλαμβάνονται στην εντολή της ενέργειας. Αλλά εδώ εμφανίζεται μία διάσταση. Πρώτον, προβλήματα εξασφάλισης της βεβαιότητας στην προμήθεια συντροφοδοσία σε φυσικό αέριο. Δεν θα υπερβάλλω, είμαι και γέρος πια. Θα σας θυμίσω ότι την εποχή της ε, γεροντοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν κακή μεν η γεροντοκρατία, αλλά τουλάχιστον την προβλέπαμε. Τώρα έχουμε μια νέα κατάσταση που θα τη χαρακτηρίζα ως σχετικώς απρόβλεπτη. Που στον τομέα της ενέργειας με το ζωτικό χαρακτήρα που διαδραματίζει δεν είναι κάτι το ε, περιθωριακό. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και αποτελεί κάτι το αρκετά ανησυχητικό. Η κρίση η ενεργειακή έρχεται μια στιγμή που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως στιγμή γενικά ηρεμίας, διότι η τιμή του πετρελαίου είχε φτάσει στο 1 τρίτο της τιμής του το καλοκαίρι. Με ανησυχεί μια τέτοια συνέπεια. Μήπως αυτό οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να ξανασυζητά θέματα που δεν ήταν ε, δεσμευμένα, που δεν ήταν δεσμεύσεις, αλλά ήταν, ψήλωση, ήταν συμφωνίες, φερειπίν, τις δεσμεύσει μας εν ώψη του 2020. Δηλαδή, με το πετρέλαιο φθηνό και την κρίση που υπάρχει και ελπίζω να μην κρατήσει πολύ, μήπως υπαναχωρήσουμε σε κάποιες δεσμεύσεις που είχαμε ε, αναλάβει έναντι της ε, θέρμανσης του κλίματος. Αυτό, αυτά όλα για να σας πω ότι τι έγινε από τη στιγμή που ξεκίνησε η εντολή μέχρι σήμερα. Κάθε ομάδα προβληματισμού θα έμπλεκε με αυτό το θέμα. Γι' αυτό ακριβώς η πρώτη συνάντησή μας ήταν χτες για να συζητήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητούμε και τι αποτελεί και τι, τι στηρίζει το πλαίσιο αυτό. Διότι Η οικονομική κρίση είναι τόσο μεγάλη που κατά την άποψή μου δεν έχει προηγούμενη. Είναι μια κρίση όπου ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει επί της διάγνωσης, των λόγων της, αν μπορούμε να μιλήσουμε για διάγνωση, και ούτε γνωρίζουμε μέχρι πού θα, ε, τι θα βρούμε μέχρι πού θα φτάσουν οι εκπλήξεις που προκύπτουν από τα διάφορα επενδυτικά ταμεία ε, που επένδυαν από εδώ και από εκεί χαμογελαστά τα τελευταία δέκα χρόνια. Στο, έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτό το σενάριο ασάφειας να θεσπίσουμε τους μέσο και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε τι δυνατότητες έχει η Ένωση για να πετύχει τους στόχους αυτούς. Εγώ λοιπόν ενώ λίγη, θα σα έλεγα μεταξύ της πρώτης συνάντηση, της συστατική συνάντηση του Δεκεμβρίου και της χθεσινή, είχα προτείνει ως πρόεδρο, μια σειρά προτεραιοτήτων που μπορώ να σας τις αναφέρω αλλά προσέθεσα και άλλες. Πρώτη προτεραιότητα κατά την άποψή μου το οικονομικό μοντέλο και το μοντέλο κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορεί να παραμείνει, να διατηρηθεί μέσα στον 21ο αιώνα. Να ξανααναλύσουμε δηλαδή την ατζέντα της Λισαβόνας ως προς το πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε μια παγκόσμια οικονομία. Ελπίζω να μην υπάρξει μια υπαναχώρηση προστατευτική στον κόσμο λόγω της κρίσης, πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε, πώς μπορεί η οικονομία μας να προσθέσει αξία, ούτω ώστε με την προστιθέμενη αξία να επανέλθει σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο που στήριξε την επιτυχία της Δυτικής Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής. Πώς μέσα σε μια οικονομική παγκοσμιοποίηση και μέσα σε έναν ανταγωνισμό ελεύθερης οικονομίας θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να προασπίζουμε ένα μοντέλο που είναι και ανταγωνιστικό και μοντέλο κοινωνική συνοχή που δεν μπορούν να διαχωριστούν. Πρώτο σημείο κατά την άποψή μου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία από τη μια και για την κοινωνική συνοχή από την άλλη. Αν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία, η βιωσιμότητα της κοινωνικής συνοχής κινδυνεύει περισσότερο από αν είχαμε ένα μοντέλο με βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και της ε, συνοχής. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη προτεραιότητα. Μπορούμε να την κόψουμε σε δύο-τρεις, ε, αλλά το είπαμε και στην ομάδα να εξετάσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι που ήθελε να κάνει και η Λισαβόνα το αποτέλεσμα 9 χρόνια μετά την ατζέντα της Λισαβόνα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητικό για κανένα στην Ευρώπη. Και πώ θα δούμε το ζήτημα τη κοινωνική συνοχή τόσο από την οπτική γωνία των εσωτερικών κρίσιμων στοιχείων, ε, δημογραφική πυραμίδα στην Ευρώπη, αλλαγές της κοινωνικής δομής τα τελευταία 40 χρόνια, μαζί με την δημογραφία δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης και τον αντίκτυπο της μετανάστευσης και άλλα, τι άλλα ενδογενή και εξωγενή στοιχεία περιλαμβάνει το κράτος πρόνοιας που πρέπει να αλλάξουμε τη στιγμή που πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα ε, πραγματικότητα. Δεύτερη προτεραιότητα. Το προηγούμενο είναι δύο ερωτήσεις. Το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης και η ικανότητα ανταγωνισμού σε μια οικονομία, ανοιχτή οικονομία, κοινωνική συνοχή Δεύτερο, ενέργεια και αλλαγή του κλίματος. Δεν θα μιλήσω πολύ γι' αυτό. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι και να τους μειώναμε στα γνωστά ως 3,20. 2020, μείωση 20% για να πετύχουμε τους στόχους υποκατάστασης ε, των, των ορυκτών καυσίμων από άλλες θα χρειαζόταν να υπάρξει να γίνει μια πραγματική επανάσταση στη χρήση των ενεργειακών πηγών, την διαφοροποίηση των δικτύων μεταφορών και των πηγών μεταφορός ενέργειας. Αυτό θα προσέφερε τεράστια ευκαιρία να προεξοφλήσουμε ως μοντέλο κάτι που βλέπουμε ότι ευτυχώς Ευτυχώς ε, υποστηρίζει η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ομπάμα παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ευτυχώς, ίσως να, είχαμε, να έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε μια μεγάλη συμμαχία για να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της ενέργειας και το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Δεύτερο πακέτο προτεραιοτήτων λοιπόν το οποίο είχα σκεφτεί να περιλάβει η εντολή Άλλο ζήτημα τώρα, οι μεταναστευτικές ροές, τόσο από την οπτική γωνία της ιδέας που έχουμε συχνά ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι πρόβλημα, όσο και από την προοπτική της αναγκαιότητας για την Ευρώπη μεταναστευτικών ροών. Λάβετε υπόψη αυτό που είπα προηγουμένως για τα δημογραφικά. Η αντίληψη της μετανάστευσης ως προβλήματος και ως ανάγκης θα πρέπει να έχει λύση. Όλος ο κόσμος το ξέρει, αλλά Δεν μπορούμε να έχουμε 15, 12, 20 μεταναστευτικέ μεταναστευτικές πολιτικές και ένα ενιαίο εσωτερικό χώρο χωρίς ε, σύνορα. Δεν μπορεί... Ε, το μόνο που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ως τοπικό είναι οι, μηχανισμοί προσαρμογής και ένταξης αυτών των μεταναστευτικών ροών αλλά να έχουμε μία μεταναστευτική πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι η ελευθερία κυκλοφορίας επηρεάζει και τη μετανάστευση. Άλλο πρόβλημα. Το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας θα ξεπεράσει την παραδοσιακή μορφή των απειλών. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα. Και άλλες απειλές θα υπάρχουν. Κάποια ε, διαλυμένα κράτη εδώ κοντά στα σύνορα της Ευρώπης κάποιες περιοχές ρήξης στον Κάφκασο, το ένα άλλο πρόβλημα στην Εγγύς και Μέση Ανατολή δίπλα στην Ευρώπη. Μην ε, σας εντυπωσιάζει το τι θα γίνει στις περιοχές αυτές του κόσμου. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να εξετάσουμε για κάποιες άλλες διαστάσεις ασφάλειας εν του 2020. Δεν θέλω να φοβήσω κανένα. Σκεφτείτε ωστόσο τι θα συμβεί αν το 2014 η ημερομηνία κατά την οποία λύγει η σύμβαση Ουκρανίας-Ρωσίας για την χρήση των ε, Ουκρανικών λιμένων από τον ε, Ρωσικό στόλο. Τι θα συμβεί αν καταγγελθεί το 2014 η, σύμβαση αυτή, η συμφωνία αυτή. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα έχει την διέξοδο αυτή στη θάλασσα. Σκεφτείτε τα. εγώ σκεφτεί και ένα πέμπτο θέμα που σχετιζόταν με τα προηγούμενα. Χρειάζεται η ευρωπαϊκή κοινότητα μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που να βαρύνει σε διεθνές επίπεδο. Θα έπρεπε στις εξωτερικές σχέσεις τώρα να προσθέσουμε το εξή. Πώς θα εκμεταλλευτούμε τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση που θα ε, αλλάξει κάτι. Μπορεί να υπερβάλλουμε ως προς αλλά κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν. Το 2005 δεν ανανεώθηκε η στρατηγική Βορειοατλαντική Συμμαχία. Το 1995, συγγνώμη. Έκτοτε άλλαξαν πολλά πράγματα. Μήπως έπρεπε να επαναξετάσουμε αυτό το στρατηγικό σχήμα. Σε δύο βασικές πτυχές τουλάχιστον. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ήδη νομίζω δέχονται ότι θα συνεχίσουν να είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο, αλλά ότι δεν μπορούν μόνες τους, μονομερός δηλαδή, να δουλεύουν, διότι η μονομερής λήψη αποφάσεων δεν είναι αποτελεσματική. Ούτε για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, ούτε η παγκόσμια κρίση ασφάλειας, ούτε για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ενέργειας ε, και της θέρμανσης του κλίματος. Οι ΙΠΑ μόνες τους δεν μπορούν. Ο νέος πρόεδρος φαίνεται ότι το καταλαβαίνει αυτό. Αν η Ευρώπη ή αν θέλετε η Αμερική, Λατινική Αμερική καταλαβαίνει πως χωρίς τις ΙΠΑ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κι εμείς. Έχουμε χώρο συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, της ενέργειας, της βελτίωσης του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Και αυτό είναι μια θέση που αναμειγνύει το άμεσο με το μεταγενέστερο. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, την, να λειτουργήσουμε σε μια πολιτική κατά της κρίσης τώρα και με μια προοπτική μελλοντική. Μπορούμε να λειτουργήσουμε μία αντικυκλική, μάλλον η αντικυκλική αντιμετώπιση της κρίσης μπορεί να, πρέπει να έχει διαστάσεις μέσω και μακροπρόθεσμες. Γι' αυτό έλεγα ότι κάποια, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποια πράγματα, ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα επηρεάσει τη στρατηγική για την ε, ενέργεια της Ευρώπης, της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλων χωρών. Διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα γυρίσουμε πίσω με πολύ επικίνδυνο τρόπο και δεν νομίζω θα μπορέσουμε να κερδίσουμε ότι χάσαμε. Διότι έχω το φόβο ότι αν ξαναρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας, που εύχομαι να είναι γρήγορη, θα ξαναυπάρξει μια κρίση ε, προμήθειας, τροφοδοσίας σε ενέργεια, επάρκειας σε ενέργεια και φτού και από την αρχή. Στην ομάδα, και αυτό είναι μια ε, πληροφορία που σας δίνω, ε, ζήτησα, μάλλον πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Και ως προς το τι είναι Ευρώπη, δηλαδή από την οπτική γωνία των συνόρων της Ευρώπης. Εγώ θα προτιμούσα να λέω τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν λέμε τι είναι η Ευρώπη πάντα μου δημιουργεί μια σημαντική αβεβαιότητα. Αν λέω τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορώ να απαντήσω εγώ, χωρίς να δεσμεύσω την ε, ομάδα, λέγοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχουν αυτοί που θέλουν να είναι μέρη μιας ομάδας χωρών της Ένωσης και πληρούν κάποιους όρους. Τώρα, το τι είναι η Ευρώπη το συζητάμε 3.000 χρόνια. Ακόμα και τώρα δεν είμαστε σίγουροι για το τι είναι. Πιστεύω ωστόσο ότι μια συζήτηση για την ταυτότητα και τις αξίες της Ευρώπης είναι σκόπιμη σε αυτή την περίοδο κρίσης. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που επιδιώκει το Κοινοβούλιο, τα θεσμικά όργανα, πολιτικοί ηγέτες και που δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα σωστό. Πώς σχετίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους πολίτες. Τι γίνεται με τους πολίτες. Ποιες είναι οι δύο διεπικοινωνίες που φεύγουν από, που βγάζουν την Ευρώπη από τη σελίτ, το στενό κύκλο και φτάνει η Ευρώπη στους πολίτες. Πότε οι πολίτες θα αισθανθούν ότι τους αφορούν οι ευρωεκλογέ που θα γίνουν σε λίγο. Όλοι γνωρίζουμε, για παράδειγμα, για τι ευρωεκλογέ ότι δεν θα τρέχουν οι πολίτε στι κάλπες στις ευρωεκλογέ. Αυτό έχει επίδραση στην Ευρώπη. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής. Δεν είμαι αξιόπιστο κατά συνέπεια. Πιστεύω στην Ευρώπη και πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του, για τον κόσμο το να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δώρον μάνεξ ουρανού. Ξέρετε, δεν είμαι πολύ πιστός γιατί κάποτε, κάποια στιγμή με εγκατέλειψε η πίστη, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι δώρο εξ ουρανού. Η, η Ευρώπη πρέπει να έχει μία εύλογη σημασία στην Ευρώπη και αυτό το επιτυγχάνει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό με ανησυχεί η αυξανόμενη αδιαφορία του Ευρωπαίου πολίτη έναντι αυτού του κοινού πεπρωμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά με ανησυχεί το γεγονός ότι πολλοί ηγέτες συμμερίζονται αυτή την απογοήτευση, αυτό το desaffectio σοκιετάτη την απομάκρυνση της κοινωνίας. Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες θέλουμε να δουλέψουμε στον, στην ομάδα, εξετάζοντας ενδεχόμενα ότι όντως η προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε, σε μελαγχολία, διότι ε, αυτό που θέλουμε επίσης είναι να ζητήσουμε την συνεισφορά όλων των ε, ενδιαφερομένων ε, δομών, Κοινοβουλίου, Επιτροπής, Ερευνητικών Οργανισμών, αλλά δεν θέλουμε η έκθεση να είναι μια εγκυκλοπαίδεια, αλλά ένα σύντομο κείμενο, 20-25 σελίδες που θα μπορούν να το διαβάσουν όλα, να, όλοι να μπορούν να το καταλάβουν. Να χρησιμοποιούμε, και δεν θέλω επίσης να χρησιμοποιούμε ε, όλες αυτά τα αρχικά που νομίζουμε ότι τα ξέρουν όλοι, αλλά δεν τα ξέρει κανένας. Κανείς πέρα έξω από το στενό κύκλο δεν ξέρει τι είναι όλα αυτά τα ε, αρχικά. Ένα κείμενο λοιπόν 25-30 σελίδων, στο οποίο μπορεί να, το οποίο μπορεί να παραπέμπει σε κάποιες συμπληρωματικές εκθέσεις. Θα θέλαμε να έχουμε έναν μόνιμο διάλογο με το Κοινοβούλιο και μέσω του Κοινοβουλίου θα θέλαμε να υπάρχει μια δυνατότητα να ανοιχτούμε και προς τους πολίτες. Εμείς ως ομάδα ούτε λεφτά έχουμε, ούτε μέσα για να ξεκινήσουμε έναν ε, ηλεκτρονικό διάλογο με τους πολίτες. Θα μπορούσε το κοινοβούλιο, όπως την εποχή της συνέλευσης, να παράσχει την υποδομή για έναν διενεργό διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες. Επαναλαμβάνω ότι δεν δεσμεύω την ομάδα προβληματισμού. Με ανησυχεί ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μέσα σε μια κρίση που δεν είναι ε, ε, επικίνδυνη ακόμα, αλλά που ε, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για να αποκτήσει Ευρώπη σημασία για τον πολίτη και για τον κόσμο. Η ευρωπαϊστική διαδέσμευση δέσμευσή μου αυξάνεται. Αν και η ανησυχία μου αυξάνεται επίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοντζάλες για την παρουσίαση αυτή των πρώτων ιδεών από την ομάδα προβληματισμού. Με μεγάλη χαρά να δεχθούμε την ε, πρόσκλησή σας να συναντηθούμε και μέσω ημών να περάσουν κάποιες ιδέες στους πολίτες. Ε, βεβαίως όπως θα ξέρετε υπήρχαν δισταγμοί για το κατά πόσον ένα βήμα σοφών ε, θα μπορούσε να κάνει μια δουλειά που ε, ήταν η δουλειά που κάνανε παλιότερα συνελεύσεις οι συνελεύσεις με συμμετοχή πολύ ευρύτερη εν πάση περιπτώσει ε, ελπίζω ε, η έκθεση όταν θα φτιαχτεί η έκθεση 2010 σε ένα χρόνο, ένα και κάτι δηλαδή από σήμερα να μην μπει στα χρονοτούλαπα η έκθεση αυτή αλλά να δημιουργήσει μια δική της δυναμική δεν αρκεί μια χρονιά ή δυο για να προχωρήσουμε στο μέλλον ε, εδώ πρόκειται για γεγαντιαίως ζητήματα και θέματα ε, πρόκειται για τη μοίρα, για το μέλλον, για το πευρωμένο της Ευρώπης δεν ξέρω πώς να το πω η ομάδα καλείται να κάνει λιγάκι τον προφήτη 2020-2030 είναι πολύ μακριά. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ε, τάσεις, οι μεγάλες τάσεις ε, που ε, ήδη από τώρα διαφαίνονται ε, από ό,τι κατάλαβα βέβαια η ομάδα είναι αρκετά αισιόδοξη ότι θα αντιμετωπίσει, θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Ε, βεβαίως ε, τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει κάποιους ε, όρους αν θέλετε ε, και χωρίς να λάβετε υπόψη σας ορισμένα πράγματα, ε, ορισμένους όρους αυτού του Ευρωπαϊκού που προήλθαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, επειδή δεν είστε πανεπιστημιακοί ή πανεπιστήμια ή φιλόσοφοι μονάχα αμφισβητών θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτές. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλοί που ζήτησαν το λόγο. Τρία λεπτά χρόνος αγόρευσης παρακαλώ. Ο πρώτος είναι ο Jean-Luc De α, ο Μέντες Τεβίγκο ήταν πιο, πιο πρώτος. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Φελίπε Γκονζάλης, πρώην συνάδελφο, παλαιότερο φίλο μου. Επίσης με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα τα όσα έχει να πει και πιστεύω ότι ε, όχι μόνο έθεσε τους σωστούς προσανατολισμούς, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι ε, κατάφερε να μεταφράσει τους προσανατολισμούς αυτούς σε κάτι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι ο χρόνος που πέρασε ανάμεσα στη στιγμή εκείνη που συστάθηκε η ομάδα προβληματισμού και σήμερα είναι ουσιαστικά ένα προνόμιο για την ομάδα αυτή. Το ότι πέρασε ο χρόνος αυτός και ότι επήλθε μάλιστα και η κρίση είναι θετικό, γιατί η κρίση νομίζω ότι έθεσε κάποια ζητήματα, μας έκανε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο την παγκοσμιοποίηση, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις της για την καθημερινή ζωή των πολιτών, καθώς επίσης και για το ρόλο που θα μπορούσε να διδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε περισσότερο συνειδητοποιημένοι μετά την κρίση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό όμω να αντιδράσουμε πια πολύ γρήγορα. Τώρα, η προοπτική που τίθεται για το 2010 θεωρώ ότι είναι θετική. Κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής που διανύουμε, συντοποιούμε κάποια πράγματα, επιστρέφουμε στη συνέχεια στην καθημερινότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αποφεληθούμε τις γνώσεις αυτής που έχουμε τώρα για να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προβληματισμοί που μας έθεσε ο Φελίπε είναι σωστοί και νομίζω ότι τους προβληματισμούς αυτούς α, συμμερίζεται και ο ίδιος ο Ευρωπαίος πολίτης. Κλιματικές αλλαγές, οικονομική κρίση, όλα αυτά απασχολούν πλέον και τον Ευρωπαίο πολίτη και συντοποιεί ο Ευρωπαίος πολίτης ότι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, οι εθνικές αρμοδιότητες δεν αρκούν πλέον, ότι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα πειράσει και την στάση του Ευρωπαίου πολίτη για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όντως ο Ευρωπαίος πολίτης πολύ συχνά δεν αισθάνεται ότι είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αισθάνεται περισσότερο πολίτης ενός κράτους μέλους. Αν όμως θέλει να διαδραματίσει τελικά ένα ρόλο στον παγκοσμιοποιημένο αυτό κόσμο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της Ευρώπης. Και η μεγάλη πρόκληση σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς να υπάρχει ένας ενθουσιασμός στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να φέρουν το ευρωπαϊκό όραμα. Δυστυχώς πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το δεδομένο. Κάτι που έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο, το οποίο όμως δεν είναι θετικό. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες πλέον θεωρούν παράλληλα ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια απειλή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Θεωρώ λοιπόν ότι για την πρόκληση αυτή η ομάδα προβληματισμού μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πρώτον η ομάδα αυτή προβληματισμού να είναι σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, να μην λειτουργήσει απομονωμένη. Και έχουμε και την εμπειρία της συντακτικής συνέλευσης, όπου είδαμε ότι αν ανοίξουμε κάπως συστήσεις μας προς τα έξω, αν εμπλέξουμε περισσότερο τον Ευρωπαίο πολίτη, τα πράγματα δεν μπορεί παρά να κινηθούν λίγο πιο θετικά. Πρώτον λοιπόν αυτόν και δεύτερον, και πάλι βασίζουμε εδώ πέρα στην εμπειρία που έχουμε από τη συνέλευση. Είναι σημαντικό προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια θετικά συμπεράσματα με την ομάδα αυτού προβληματισμού Σαφώς θα πρέπει να συνταχθεί μια έκθεση, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Μέσω της συνέλευσης, μέσω των συζητήσεων της συνέλευσης, καταλήξαμε σε ένα σύνταγμα και το σύνταγμα αυτό θα μπορούσε στη συνέχεια, εφόσον βέβαια το είχαν εγκρίνει όλα τα κράτη-μέλη, να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν και το πόρισμα της ομάδας προβληματισμού να αποτελέσει κάτι το έμπρακτο το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, να μην είναι μια έκθεση που θα μείνει κλεισμένη σε κάποιο γραφείο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τον κύριο μιλήσετε λίγο παραπάνω από τρία λεπτά Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε Γκονσάλε. Χαιρόμαστε που είστε εδώ και πρέπει να σα συγχαρούμε για την πρώτη παρέμβασή σα. Ήταν πολύ ε, ενδιαφέρουσα ε, η πρόταση που κάνετε για τις νέες σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας, τη ζωή μας και αυτή είναι μία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η σχέση αυτή μπορεί να περιλάβει και τα στοιχεία της ε, ασφάλειας. Δεν μπορεί όπως αναφέρθηκε εδώ η Ευρώπη να πληρώνει τις δαπάνες αλλά στα θέματα ε, άμυνας και ασφάλειας να μιλάμε μόνο θεσμικά και να μην εξετάζουμε τι θέλει η Ευρώπη ως σύστημα ασφάλειας. Και αυτό το λένε όλες οι έρευνες. Όλες οι έρευνες δίνουν, λένε ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντικό το ζήτημα αυτό. Δεύτερο θέμα, κλιματική αλλαγή. Ε, υπάρχει ένα θέμα που είναι ταμπού σε πολλά κράτη, που δεν πρέπει να παραμείνει ταμπού πυρηνική ενέργεια. Εμεί γενικά πρέπει να ξεφορτωνόμαστε τραμπού. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό ω μια αναγκαιότητα για το μέλλον τη Ευρώπη, ιδίω σε μια στιγμή που βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από άλλου εξωτερικού εταίρου που δεν συμμερίζονται τι ίδιε προτεραιότητε με εμά του Ευρωπαίου. Δύο σχόλια επίση. Για την ταυτότητα, μην ε, ασχοληθείτε πολύ. Εγώ χρόνια παλεύω για τα θέματα της ταυτότητας και εν τέλει σας λέω ότι δεν ε, δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχει ένας ποιητής που λέει είμαστε αυτοί που είμαστε. Το ποιοι είμαστε εμείς το ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, ε κάναμε λάθος όταν γράψαμε ότι θέλαμε να βάλουμε στη συνθήκη την αναφορά στον, στις χριστιανικές ε, αρχές της Ένωσης. Ε, είπατε ότι μερικέ φορέ οι σκέψει σα οδηγούν σε μελαγχολία. Μην το πιστεύετε αυτό. Κάθε δουλειά που κάνετε είναι χρήσιμη και δεν θα σα οδηγήσει σε μελαγχολία η δουλειά αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Euh, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ λέει κύριε Σαλέμ Γαμασούρ. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε εδώ και πάλι τον κύριο Φελίπε Γκοντζάλες και τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποστηρίζει την ε, ευρωπαϊστική του θέση. Θα πω μερικά πράγματα για να σας βοηθήσω κύριε. Πρώτον, πριν από 20 χρόνια εξελέγει ως Ευρωβουλευτής. Επί 19 χρόνια αγωνιστικά να καταλάβω ότι η, Ευρωπαϊ... το Ευρωπαϊκή νόμη που ε, ε, περνάμε για να βοηθήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη οι ευρωπαϊκοί νόμοι αυτοί δεν λειτουργούν καλά για τις επιχειρήσεις λειτουργούν για την η αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων η, ε, αποζημίωση σε θέματα ιατρικής περίθαλψης, η ελευθερία εγκατάστασης, η ε, ελευθερία η μεικτή γάμη και δεν ξέρω τι. Αυτά όμως δεν λειτουργούν για σε οικονομικό επίπεδο και επιχειρησιακό, επιχειρηματικό επίπεδο μπορεί κάποιοι, κάποιοι νόμοι να λειτουργούν. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει στην προσέγγιση των πολιτών. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι πρέπει να μην υπάρχουν σύνορα κτλ. κτλ. Όμως στα σχολιά μας όλοι φτιάχνουμε εθνικιστές σε όλες τις περιφέρειες μας, σε όλες τις, σχολέ, χώρες διδάσκουμε τα παιδιά μας την ιστορία, την εθνική που είναι στεφανωμένη με δόξα και θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ε, δοξασμένη αν είχαμε ε, κάνει ε, πολέμους με τους γειτονές μας και τους είχαμε νικήσει. Λοιπόν, γιατί στη διδασκαλία της ιστορίας δεν υπάρχει αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτο θέμα, ευρώ, ενιαίο νόμισμα. Εντάξει, κάποια επιτυχία είναι ε, ε, την περασμένη εβδομάδα το γιορτάσαμε όμως αυτά έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο που πρέπει να αναρωτηθούμε μας συμφέρει να συνεχίσουμε με το ευρώ για να φτιάξουμε ένα μεγάλο ευρώ ανταγωνιστή του δολαρίου ή, θα ήταν καλύτερα προς το συμφέρον να διατηρήσουμε ως ευρωπαϊκό και μόνο νόμισμα το ευρώ και όχι να το κάνουμε παγκόσμιο Τέταρτο θέμα, η πολιτική γειτονία. Επα, την επανεφίβραμε σε σχέση με τις γειτονικές χώρες δεν μπορούμε ε, να ε, τους πούμε να γίνουν κράτη-μέλη της Ένωσης αλλά θέλουμε καλές σχέσεις, ειρηνικές σχέσεις μεταξύ τους και με εμάς και τα λοιπά θέλουμε να είναι δημοκρατίες και από εκεί και πέρα οι χώρες αυτές είναι οι χώρες γειτονίας που λέμε ε, τι ε, πρέπει να σκεφτούμε όμως καλύτερα τη σχέση και το τι θέλουμε από τις χώρες αυτές επόμενο θέμα την παγκοσμιοποίηση εδώ του 21ου αιώνα. Είμαστε παράδειγμα γιατί. Είμαστε παράδειγμα για ε, μια ένωση χωρών που γειτονεύουν. Υπάρχει όμως η, το Μερκοσούρ, υπάρχει οι χώρες του κόλπου, υπάρχει η Αφρική και η ε, και Ένωση κτλ υπάρχουν λοιπόν και ε, άλλοι οργανισμοί χωρών. Εμείς είμαστε ένας από αυτούς. Ε, δεν θα μπορούσαμε εμείς να εμπνευστούμε από αυτά που κάνουν άλλοι οργανισμοί, άλλοι ομάδες, άλλες ομάδες χωρών. Ε, ο κύριος Λαμασούρ λέει ο πρόεδρος όπως και οι παλιοί ε, πρωθυπουργοί, οι τέος πρωθυπουργοί έχει πολύ καλές ιδέες. Ο κύριος Σαβαρά θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που μας είπατε και να αναφέρω και κάποιες άλλες ιδέες. Λοιπόν, όπως είπατε, ε, έχουμε τη διάγνωση, έχουμε και τη θεραπεία. Καλά, αλλά το κόστος της θεραπείας ή της εντατικοποίησης της θεραπείας ποιο είναι. Μπορεί αν δεν ενισχύσουμε αν θέλετε τη θεραπεία το κόστος να είναι μεγαλύτερο από ότι αν την ενισχύαμε. Δεύτερο θέμα. Διανύουμε κρίσεις. Κάποιες κρίσεις είναι έκτακτες ευκαιριακές και κάποιες άλλες διαρθρωτικές. Εμείς εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις διαρθρωτικές κρίσεις και όχι τις περιστασιακές. Τρίτο θέμα αναφερθήκατε στην ταυτότητα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Εμείς, εγώ νομίζω ότι και εδώ υπάρχει κρίση και μιλάμε για διαρθρωτική κρίση. Ε. Έχουμε κρίση ταυτότητας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Α, δεν εννοώ να το δούμε τα φυσικά βεβαίως το θέμα αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα ή ένα όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που να μπορέσει να κινητοποιήσει τους πολίτες και θα πρέπει να ορίσουμε και τα κριτήρια της συνοχής γιατί αυτά τα κριτήρια είναι αυτά που προσδιορίζουν το γιατί ο πολίτης πρέπει να είναι πιστός στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στα ευρωπαϊκά όργανα. Και οι βασικές λέξεις είναι ασφάλεια με την έννοια της security ατομική, συλλογική, πολιτιστική και διεθνής. Security όμως, ασφάλεια έτσι. Εάν και στο, σε κάποια από τα θέματα αυτά η, η, Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να, προσθέ, να, να, να, φτιάξει μια προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτό που παρέχουν τα ε, εθνικά κράτη τότε είμαστε δεν χρειάζεται να ζητούμε τίποτα άλλο. Επόμενη ιδέα. Θεωρούμε ότι τα εθνικά κράτη, θεωρείται ότι τα εθνικά κράτη απειλούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την ενοποίηση αν θέλετε της Ευρώπης. Ο κατακαιρματισμός των εθνικών κρατών, η αναρχία που κυριαρχεί σε κάποια κράτη μέλη όπου ο πολίτης αισθάνεται πιο ασφαλής στις, σε μικρότερες ομάδες οι οποίες όμως είναι λιγότερο ελεύθερες αυτό είναι το πρόβλημα του Ευρωπαίου πολίτη εγώ δεν είμαι τέος πρωθυπουργός λέει ο μιλήτης είμαι τέος αντιπρόεδρος κυβέρνησης, δώστε μου και εμένα κανένα λεπτάκι επιπλέον. Ναι, θέλω να πηχήσω κλείνοντας αυτά που είπε ο Λέων Λαμασούρ. Πώς θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα με εθνικούς όμως αρχιτέκτονες. Έτσι, ε, δεν είναι δυνατόν να δεχθεί να δεχθούν ε, δεν μπορούν οι εθνικοί αρχιτέκτονες να δεχθούν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ευρωπαϊκό όραμα. Χρειαζόμαστε Ευρωπαίους αρχιτέκτονες λοιπόν. Και κλείνοντας λέω ότι θα πρέπει να φτιαχτεί ένα πολιτικό μανιφέστο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Ένα τεχνικό πρόγραμμα δράσης που να μπορούν να το καταλάβουν και οι πολιτικοί και οι τεχνοκράτες και οι πολίτες. Μαρία Στέβε, Μάριο Στέβες δεν είστε όμως τέος πρωθυπουργός, είστε μέλλον. Τέλο πάντων, εντάξει, άντε τότε σας δώσουμε πέντε λεφτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχάς αυτή την ομάδα προβληματισμού γιατί πραγματικά την έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι όντως αυτή η ομάδα προβληματισμού θα καταφέρει να θέσει τους προσανατολισμούς για το μέλλον. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα πιο συγκεκριμένα στην παρέμβαση του κυρίου Κοντζάλης. και θα ήθελα να κάνω κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις, όχι επικρίσεις στην ε, παρουσίασή του. Σαφώς υπάρχει το πρόβλημα της κρίσης και η μη προβλεψιμότητα της κρίσης αυτής. Αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο αβέβαιο και καταλαβαίνετε ότι μπορεί μόνο να βρεθεί ή πρέπει να βρεθεί μια παγκόσμια κοινή λύση στην ε, συστημική κρίση που αντιμετωπίζουμε και θα αποτελέσει αυτό το πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί και μια παγκόσμια δικαιοσύνη, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Πρέπει λοιπόν η ομάδα προβληματισμού να καταφέρει να θεσπίσει ένα τέτοιο μοντέλο, ένα μοντέλο που θα επιφέρει μια λύση στην κρίση αυτή. Να δούμε στα πλαίσια του μοντέλου αυτού πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα καταφέρουμε να οριοθετήσουμε τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιοι είναι οι περιορισμοί και τα όρια της Επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα καταφέρουμε να εξαγάγουμε στο εξωτερικό στη συνέχεια το μοντέλο αυτό. Αν ε, εξετάσουμε την περίοδο 2020-2030 θα μπορούσαμε σαφώς να είμαστε οραματιστές και να επικεντρωθούμε μόνο τελικά στο παρελθόν και να αναφερθούμε στην περίοδο του διαφωτισμού λέγοντας ότι η παγκόσμια αυτή δικαιοσύνη μπορεί να έρθει μόνο μέσω μιας ένωσης των ε, λαών, ότι ε, η παγκόσμια αυτή δικαιοσύνη μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ε, συμβολής των φιλοσόφων, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα, τα οικονομικά, τα μοντέλα των διεθνών σχέσεων και ότι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η ακόλουθη. Η ομάδα αυτή πώς θα ορίσει τελικά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίως και πώς θα καθορίσει τελικά τις μελλοντικές δυνατότητες διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρει να δημιουργήσει μία παγκόσμια δικαιοσύνη και πώς θα μπορούσε τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας χώρος μεστός ταυτότητας και όχι ένας χώρος όπου αποσιάζει τελικά η ταυτότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα τεράστιες δυνατότητες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Ευχαριστώ. Κάρλος Κανέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κονζάλης μας είπε ότι αντιμετωπίζουμε μια θεσμική κρίση. Θεωρώ όμως ότι η κρίση αυτή είναι πολύ πιο βαθιά. Πρόκειται για μια σταγματική κρίση, όχι επειδή δεν επικυρώθηκε το Σύνταγμα. Το θέμα δεν έχει να κάνει με τη διαδικασία, δεν είναι διαδικαστικό, έχει να κάνει με την ίδια τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ε, κυβερνήσεων λαού έχει να κάνει με την πραγματική την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, έχει να κάνει ουσιαστικά με την κρίση εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορείτε να φανταστείτε να υφίσταται τελικά ένας πολιτικός οργανισμός εν μέσω της κρίσης αυτής χωρίς τον κίνδυνο να καταρρεύσει. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση της κρίσης επίσης και στις επόμενες εκλογές, στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. κινδυνεύουμε δεχομένω να οπισθοδρομήσουμε και να καταλήξουμε τελικά σε ένα κενό. Και οι πολίτες τελικά θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι χρήσιμη η παρουσία μας. Τώρα, ποια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα σας. Στο Σύνταγμα υπάρχει ένα άγραφο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να προβλεφθούν όμως οι κατάλληλες διαδικασίες και οι κατάλληλοι θεσμοί προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε στις πολιτικές αυτές οικονομική και κοινωνική πολιτική. Νομίζω ότι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε μια ουσιαστική οικονομική πολιτική με την υποστήριξη των κυβερνήσεων. Και αρκούν τελικά μόνο οι ευρωπαϊκές εκλογές για να ακουστεί η φωνή του λαού. Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες δύο διαβούλευσεις πέρα δηλαδή από τα δημοψηφίσματα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα επόμενα 20-30 χρόνια αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές οι οποίες δεν είναι καθαρά θεσμικές, είναι συνταγματικές κατά την άποψή μου. Πρέπει δηλαδή να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εμπλέξουμε ως το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τα δίκτυα αυτά που θα μας επιτρέψουν μια καλύτερη διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά. Πολύ ωραία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο για τις μεγάλες τάσεις στην Ευρώπη και υπήρχε στην αρχή μία εικόνα για το 2025 όπου ο David Beckham, πρόεδρος της Ευρώπης, δέχεται τον, τον Κινέζο αυτοκράτορα και τον ευχαριστεί γιατί τελικά βοήθησαν πάρα πολύ στο να σωθεί η Βενετία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς να περιγράφει το μέλλον. Αν όντω έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, σας εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία. Νομίζω πάντως ότι ακούσαμε ήδη μία πολύ θετική προσέγγιση από τον κύριο Γκοντζάλες. Εσείς είπατε κύριε Γκοντζάλες ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην επικαιρότητα και στις υφιστάμενες συνθήκες, αλλά στους ε, όρους εκείνους που θα μας επιτρέψουν να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα χρονικό ορίζοντα 2020, 2025, 2030. Πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πριν από μισό χρόνο αυτό το οποίο μας απασχολούσε περισσότερο ήταν η αύξηση των τιμών των τροφίμων. Τώρα βλέπουμε ότι καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε άλλα διαφορετικά προβλήματα. Συνεπώς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε πάντα προσεκτικοί και να κατευθύνουμε τελικά την προσοχή μας στους παράγοντες εκείνους που θα καθορίσουν, που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Και ήδη εσείς αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και το πιο ουσιαστικό ζήτημα προκειμένου να καταφέρουμε να κερδίσουμε τον αγώνα της Ευρώπης, γιατί δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να σχεδιάσουμε το μέλλον αν έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη. Και όπως ε, είπατε κι εσείς, στο ζήτημα αυτό διανύουμε μια κρίση. Τώρα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών. Πρώτον, πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουν πλέον οι θεσμικές συζητήσεις. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτές. Σαφώς είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Τώρα πρέπει όμως να τελειώσει πια η συζήτηση και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη συζήτηση αυτή και να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Α ολοκληρωθούν οι συζητήσει αυτές και ας μην απασχολούμε τους πολίτες με τις συζητήσει αυτές γιατί απλώς δεν ενδιαφέρονται. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ενδεχομένως να μας ευχαριστεί κιόλα, αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τόσο πολύ τον Ευρωπαίο πολίτη. Δεύτερον, ταυτότητα η ταυτότητά μας ε, έχει να κάνει ουσιαστικά με το τι μας έχει κληροδοτηθεί, ποιο είναι το ευρωπαϊκό κληρονόμημα. Αναφερθήκαμε, κληροδότημα με συγχωρείτε, αναφερθήκαμε, αναφερθήκε κάποιος στις χριστιανικές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πράγματα. Οι ίδιοι πολίτες, οι πρωτοβουλίες των πολιτών αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επομένως, θα πρέπει βάσει αυτών να καθορίσουμε και το μέλλον της Ευρώπης, να βασιστούμε σε αυτούς τους παράγοντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καβόσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την παρέμβαση που έκανε και την ανάλυση που έκανε της κατάστασης. Θα ήθελα να προσθέσω μια νότα αισιοδοξία στην απεσιόδοξη εικόνα που μας έδωσε για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη. Στο πανεπιστήμιο όπου δουλεύω έγινε ένα διαγώνισμα μεταξύ των φοιτητών. Τους ζητήσαμε να γράψουν μια έκθεση για το πώς θα είναι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλω να πω ότι οι ιδέες τους και οι πίστη που έχουν, ε, φαίνεται να έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πραγματικά πηγή έμπνευση. Ε, βεβαίω και πραγματικά νομίζω ότι μπορεί κανείς να βρει πολίτες τους οποίους να ρωτήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η απάντηση που θα πάρει να μην είναι απεσιόδοξη. Εξαρτάται βεβαίως από τις προσδοκίες που έχει κανείς από την Ευρώπη και εξαρτάται και εδώ μιλ... μπορούμε να πούμε και μερικά λόγια τις προσδοκίες που έχουμε από την ομάδα προβληματισμού ναι, απαρτίζεται από ορισμένα άτομα η ομάδα ε, προβληματισμού που δεν είναι σοφοί μπορεί να είναι αλλά δεν είναι γιατροί να έχουν στη διάθεσή τους κάποια πανάκια για όλα τα προβλήματα. Εμείς, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή μπορεί να κάνει πολύ σημαντική δουλειά ε, και είναι και μπορεί κάλλιστα να ε, κάνει μια ανάλυση του πώς θα θέλαμε να είναι η Ευρώπη ε, σε 10-20 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε την ταυτότητά μας. Τι εστί ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Έχουμε 27 διαφορετικά ε, κράτη-μέλη με τα δικά του χαρακτηριστικά του καθένα. Η διαφορετικότητα είναι κάτι που χαιρετίζουμε. Εκείνο λοιπόν που έχει να κάνει η ομάδα ε, προβληματισμού είναι να δει τα θέματα λιγάκι πιο αισιόδοξα λιγάκι πιο θετικά γιατί για να ψάχνει διαφορές μεταξύ των 27 να ψάχνει κοινά σημεία μεταξύ των 27 και να βρείτε λοιπόν τα σημεία με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί ο Ευρωπαίος πολίτης και τα οποία είναι κοινά για όλους. ο προσδιορισμός της ευρωπαϊκής ταυτότητας ο προσδιορισμός των, στοιχείων εκείνων που μας ενώνουν ε, είναι η αρχή της δουλειάς που πρέπει να κάνετε κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βλαβεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω και σας λυπάμαι ε, το πρόβλημα που έχετε. Πολλές ερωτήσεις σας στέθηκαν πάρα πολύ προβληματικές. Δύο θέματα θέλω να θέσω. Πρώτον, ευρωπαϊκή ηθαγένεια ή αν θέλετε μια άλλη διάσταση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η δημοκρατία δημιουργήθηκε στα εθνικά κράτη. Μήπως πιστεύετε ότι πρέπει η ομάδα προβληματισμού σας να έχει ως σημαντικό αντικείμενο το πώς θα αναπτυχθεί ο χώρος δημόσιου διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καλυφθούν οι, απο, αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολίτη ε, ο οποίος δέχεται την Ευρώπη, την χρειάζεται την Ευρώπη αλλά δεν αισθάνεται ενημερωμένος και υπεύθυνο εναντί της. Πρώτη λοιπόν πρόκληση. Πώς θα δημιουργήσουμε μια στρατηγική για ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Δεύτερο θέμα. Μήπως η ομάδα θα έπρεπε να εξετάσει το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Όπως ξέρετε το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα ανάπτυξης αλλά και ισορροπίας. Υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι λευκοί πανόλης, η δημογραφική αδυναμία μας. Σε 15-20 χρόνια θα έχουμε το άχθος ενός μεγάλου αριθμού ηλικιωμένων παθητικών, αυτό το παθητικό. Το ερώτημα είναι πώς θα προετοιμάσουμε την κοινωνία πώς θα επιτρέψουμε όχι μόνο την αλλαγή της οικογενειακής συμπεριφοράς, αλλά πώς θα κατατήσουμε τους ηλικιωμένους να είναι πιο δραστήριοι, να αναλάβουν με περισσότερες ευθύνες, να τους δείξουμε ότι είναι ικανοί να δουλέψουν και να περιορίσουμε την πρόκληση της μετανάστευσης που δεν είναι αναποφευκτή. Ευχαριστώ. Θα έπρεπε να είχα κλείσει νωρίτερα τον κατάλογο των αγοριτών γιατί όλο ένα και περισσότεροι ε, ομιλητές εμφανίζονται. Μπορώ να δεχθώ όλους τους επιπρόσθετους αν μιλήσετε δύο λεπτά. Η κυρία Γεντεμέκη ε, κατόπιν. Θα μιλήσω φιλανδικά. Tehtävänne on erittäin haastava. Täällä on puhuttu... Ε, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η δουλειά που κάνετε. Μιλήσατε για τον Ομπάμα και πώς οι αποφάσεις του Ομπάμα θα επηρεάσουν την Ευρώπη και τις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Όμως η δουλειά σας είναι να εξετάσετε την προοπτική σε 10, 20 χρόνια, το 2020, το 2030. Μπορεί λοιπόν και να είναι πρόεδρος ο Ομπάμα για δύο τετραετίες, πάλι θα πρέπει να δείτε, να εξετάσετε τον αντίκτυπο των πολιτικών του μετά, στο, στο απότερο μέλλον. Άρα πρέπει να έχετε μια γενική επισκόπηση της κατάστασης εδώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να βρείτε μια λύση στο θέμα της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να έχουμε γρηγορό ε, ανταγωνισμό ταχύτερα με παράλληλα κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να βρούμε μία λύση. Αλλιώς θα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτης και δεύτερης ε, κατηγορίας. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Θα ήλπιζα να δείτε και τα θεσμικά ζητήματα, αλλά κυρίως και αυτά που πρέπει να δούμε τι περιλαμβάνει και η δική μας εντολή, όχι μόνο τα θεσμικά ζητήματα. Τα κοινά ευρωπαϊκά θέματα και να ξέρουμε τι είναι εθνική και τι είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λύση του 1930 στα προβλήματα του 1950. Αν ξαναρχίζαμε από το μηδέν τώρα φαντάζομαι δεν θα δημιουργεί το καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εδώ καθόμαστε και κουβεντιάζουμε πώς θα μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 20 χρόνια ζούμε σε μια ε, κοινωνία που τρέχει με αστρονομική ταχύτητα που τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε τα πράγματα γρήγορα τρέχουμε οι κυβερνήσεις εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να βγουν από τη μέση για να μπορέσουμε να τρέξουμε να δώσουν μια κάποια ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κοινωνία που τρέχει δεν θέλουμε περιορισμούς ή ελέγχους που μας επιβραδινούν. ήδη πολλοί από εσά αποδέχτηκαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χάνει την επαφή της με, τον πολίτη, τους πολίτες και η κρίση που διανύουμε επιδεινώνεται από κάποιες ενέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, τηρείται ο, ο, ο πρώτος κανόνας για τις πολιτικές τρύπες που λέει ότι όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια από αυτές σταματάς να σκάβεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ε, θα εξαφανιστεί ε, τα επόμενα χρόνια και δεν πρόκειται να επιζήσει μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Αυτό καταστροφική είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο πρόεδρος. Πω, πω, πω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκονζάλη και όλους τους ε, συμμετέχοντες. Αντικαθιστώ τον κύριο Μπάχαρ, τον Πρωθυπουργό της ε, Σλοβενίας, θα, ήθελα να κάνω μια παρέμβαση ε, τριών λεπτών και να κάνω ένα ερώτημα προς τον κύριο Γκονζάλες. Έχουμε την περίφημη κρίση του φυσικού αερίου. Η κρίση αυτή μας δείχνει ότι χρειαζόμαστε μια σταθερή εταιρική σχέση με την ε, Ρωσία. Σαφώς επίσης και με τις χώρες διαμεσολαβητές όπως η Ουκρανία, αλλά κυρίως με τη Ρωσία. Και το ερώτημά μου τώρα Το σχέδιο αυτό του να δημιουργηθεί μία αντιπυραυλική ασπίδα στην Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν αντιβαίνει ουσιαστικά σε αυτήν σχέση. Και το σχέδιο αυτό συμμορφώνεται τελικά με την επιθυμία του Ευρωπαίου πολίτη να είναι ασφαλής στο μέλλον. Χθες ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Τσεχίας, ο οποίος περιέγραψε το σχέδιο αυτό σε ένα σχέδιο το οποίο τελικά επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι εξημών θεωρούμε ότι το αντίθετο συμβαίνει. Η ασπίδα αυτή αποτελεί τελικά μία απειλή, γιατί τελικά ενθαρρύνει την Ρωσία να ε, μπει σε έναν ανταγωνισμό ε, εξοπλισμών. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί λίγο περισσότερο την στρατηγική και την θέση την οποία θα αναλάβει στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ιδίως με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει και σε αυτά τα ζητήματα να απαντήσει η ομάδα προβληματισμού. Σας ευχαριστώ. Ε, να απαντήσω εντάχει στα σχόλια του κ. Νταχάν όταν μίλησε τις μεγάλες επιτυχίες της συνέλευσης και να του υπενθυμίσω ότι το κείμενο που προετοίμασε η Συνέλευση απορρίφθηκε ξεκάθαρα και στη Γαλλία και στην Ολλανδία ενώ ένα αντίστοιχο σχεδόν, παρόμοιο σχεδόν κείμενο απορρίφθηκε ομοίως και στην Ιρλανδία. Δεν είναι και πολύ επιτυχημένο το κείμενο. Τώρα, για αυτά που είπε ο κύριος Γκοντζάλεφ, όταν δούλευα για το Readers Digest είχαμε περιπλανόμενους ε, εκδότες κάποιοι λέγαμε ε, έκαναν ε, έκδοση κάποιοι απλά έκαναν βόλτες περιπλανούνταν έχω την εντύπωση ότι κάποια από τα μέλη μόνο ε, σκέφτονται δεν θέλω να είμαι αγενής προς τον κύριο Γκονζάλες, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε 10 χρόνια στο κοινοβούλιο δεν άκουσα κάποιον να μιλάει 40 λεπτά χωρίς καθόλου περιεχόμενο. Έλεγε, έλεγε, έλεγε κοινότοπα πράγματα, κλεισέ, χωρίς ουσία, χωρίς πορεία, χωρίς, ε, έρμο, ε, χωρίς καμία σκέψη. Η μία ερώτηση που έθεσε ο κύριος Γκοζάλες και που συνέ, συνόψισε και τη συζήτηση και την ομιλία του είναι πώς μπορούμε να γίνουμε σημαντικοί για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολλοί το είπαν αυτό. Σημείωσα πώς προσθέτουμε αξία στους Ευρωπαίους πολίτες, πώς ξαναποκτούμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό όνειρο, γινόμαστε, απελ, απελπιζόμαστε. Τι είμαστε στα ελληνικά, στα αγγλικά, η ερώτηση είναι γιατί υπάρχει Ευρώπη και η απάντηση είναι δεν έχουμε απάντηση. Αν πάω στο δρόμο σε, σε μια πόλη του East Midlands και του ρωτήσω γιατί υπάρχει Ευρώπη, ε, δεν θα πάρουμε και πολύ ουσιαστικέ απαντήσει. Μια σειρά καταγγελιών, παραπώνων, γκρίνια, το κόστο, ε, οι κανονισμοί που μπλοκάρουν και δυσκολεύουν τα πράγματα, ότι ε, χαράμε τις παλιές μορφές ε, θερμομέτρου, τα, ε, τα παλιά που ξέραμε και υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο θέλουμε να το εξάγουμε αλλού. Ξανασκεφτείτε γιατί υπάρχετε πριν αποφασίσετε για το που θέλετε να πάτε. Ευχαριστώ κύριε Χέλμερ. Ο κύριος Γκονζάλης πρέπει να φύγει σε 10 λεπτά. Ένα λεπτό οι υπόλοιποι και μετά θα μιλήσει για λίγο ο κύριος Μπαρον Κρέσπο. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ επιτρέψτε μου να πω ορισμένα πράγματα ίσως επικριτικά. Ε, πραγματικά ορισμένα πράγματα ε, με ενοχλούν στην Ευρώπη, ε, κάπου με απελπίζουν. Η ομάδα προβληματισμού τι ε, ψάχνει, ψάχνει να βρει ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης γιατί ούτω ώστε να διορθώσει ενδεχομένως κάποια πορεία αν το κάποιες επιτροπές, κάποιες τάσεις αν τα πράγματα δεν φαίνονται να πηγαίνουν προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι μία ερμηνεία. Αν όμως προσπαθείτε να βρείτε ποιο είναι το μέλλον για να δείτε πως θέλουμε να, ζούμε στο μέλλον αν αυτή είναι η δουλειά που προσπαθείτε να κάνετε το ερώτημα είναι το άλλο μπορείτε να επιβάλλετε πως θέλουν να ζήσουν οι πολίτες της Υπήρου αυτής Οπότε, η συμπερίπτωση, το πρόβλημα δεν είναι διάλογος με τους πολίτες το πρόβλημα είναι κυβέρνηση του λαού για το λαό μέσω του λαού κύριε Πρωθυπουργέ και αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο Πρόεδρος ζητώ συγγνώμη ε, που σας περιορίζω στο ένα λεπτό αλλά τι να κάνουμε κοιτάξτε ε, εγώ νομίζω ότι εκείνο περί το οποίο πρόκειται είναι ότι να, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη και να γίνει, για να γίνει αυτό ε, Νομίζω ότι είναι σημαντικά δύο πράγματα. Πρώτον να υπάρχει ένα ενιαίο όραμα και δεύτερον να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση. Οι κρίσεις που αναφέρατε είναι η ευκαιρία που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη να συνδυάσει το όραμα και την προσπάθεια ή την ε, επίδοση αν θέλετε σε ορισμένα πράγματα. η την ε, επιδοση αν θελετε σε ορισμενα πραγματα α, εφόσον διανύουμε αυτή τη στιγμή κάποιες κρίσεις ε, η, το ευρωπαϊκό όραμα μπορούμε να το διατηρήσουμε μ, δουλεύοντας όλοι μαζί για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτού του οράματος. Ε, Ένα λεπτό λέει ο κύριος Χάν. Ο κύριος Μπαρον Κρέσπο, ε, μίλησες πρόεδρε για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και θέλω να υπενθυμίσω ότι εσύ ε, στο το αίτημα του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθεί η Ιθαγένεια στη συνθήκη του Μάστρεχτ και το πέρασε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Ζήτησε να δουλεύουμε με το Κοινοβούλιο. Ο Ντεάν απάντησε με την εμπειρία του από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος Λάινεν τώρα θα πρέπει να δει πω θα το οργανώσουμε αυτό. Κατόπιν, μια παρατήρηση. Δεν πιστεύω ότι απαγορεύεται από την εντολή του Συμβουλίου να κάνεις κάποια εύλογη πρόταση για να λειτουργήσουμε καλύτερα χωρίς να αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτά τα όλα ευχαριστώ. Merci Πολύ σύντομος. Πολλές ιδέες, σκέψεις, εν Δύσκολα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και τηλεγραφικά. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι όταν θέτουμε ερωτήματα για να μπούμε και πρέπει να μπούμε σε θεσμικά θέματα, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του Συμβουλίου μου ζήτησαν να ασχοληθούμε με την επικουρικότητα που εξορισμού δημιουργεί θεσμικά προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι αναγκαίο, πραγματικά το πιστεύω αυτό, να μιλήσουμε για την επικουρικότητα. έχουμε μια κάποια δυνατότητα να ε, παρακάμψουμε τις εντολές τους, ε, τους, του Συμβουλίου, αλλά η Ευρώπη μπορεί να αποκτήσει πιο ευέλικτα εργαλεία στα επόμενα χρόνια. Αυτό επαναλαμβάνω ωστόσο είναι προσωπική άποψη. Μπορεί και παραμένει προσωπική κρίση, η προσωπική άποψη. Η οικονομική κρίση είναι μια καλή ευκαιρία γιατί έδωσε, ανέδειξε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίση αυτή καθ' ούτε πολύ λιγότερο ότι θα εξαφανιστεί σε 10-20 χρόνια, αλλά να σας πω ότι και να υπήρχε κρίση στην Ένωση θα την ξαναδημιουργούσαμε ως μια αναγκαιότητα. Κατά πάσα πιθανότητα οι πολίτες θα, αντι, θα αν τους έλειπε αυτό που έχουν. Αυτή τη στιγμή τη δουν Εάν θεωρούσαν ότι κάτι τους έλειπε στην, στο σπίτι τους, στον οίκο τους, θα είχαμε μια νέα ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ βλέπω την κρίση ως ευκαιρία να θεωρήσεις κάποιων διαφορετικών προβλημάτων, όχι μόνο συγκυριακών προβλημάτων, διότι πιστεύω ότι η κρίση αγγίζει τη δομή της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και τη λειτουργία της διεθνούς ασφάλειας. Τι θα ήθελε λοιπόν να κάνει η ομάδα εργασία για να είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό που έκανε ε, μία επιτροπή 4-5 ατόμων με δύο συστάσεις σε δύο σελίδες όταν τους είχαν ζητήσει να ε, παρουσιάσουν τα προβλήματα, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ε, κοινωνίας της πληροφορίας. Δύο σελίδες, 12 προτάσεις. Αυτό είχε γίνει στην Ινδία. Η κυβέρνηση δεν το εφάρμοσε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την... Ε, αλλά πέτυχε διάφορα πράγματα στην ε, αντιμετώπιση της κοινωνίας της πληροφορίας από τη χώρα. Θα μπορούσαμε στο διάλογο να, αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, να συμπεριλάβουμε μία επικοινωνία με την κοινωνία της ομάδας διαμεσολάβησης. Πέραν αυτού ωστόσο θα πρέπει να δεχθούμε ότι θα υπάρξει διάλογος με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, τόσο ώστε να έχουμε επικοινωνία με τον πολίτη. Η έκθεση, έτσι όπως ε, τη σκεφτήκαμε, είναι αναφορά, έκθεση, δηλαδή το κείμενο και συστάσεις. Να πω στον κύριο Μέντες Δεβίγκο ότι η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πώς να μην περιλαμβάνει τα θέματα της άμυνας και ασφάλειας. Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο στρατιωτικοί, στο στρατό. Θα μπορούσαν το 10% από αυτόν, 150.000, να ε, δουλέψουν σαν στρατό της Ένωσης για ειρηνευτικές διαδικασίες, ό,τι θέλετε. Αλλά προφανώς η, η έννοια της υπεράσπισης του εθνικού εδάφους έχει χάσει ε, νόημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα δεν περισσότερο θα χάσει με την προστατευτική ασπίδα. Αλλά θεωρητικά αυτή η προστατευτική ασπίδα, αντιπυραυλική ασπίδα, ε, υποτίθεται ότι μας προστατεύει από την απειλή του Ιράν. Αυτό δεν το λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη, αλλά οι περισσότερο, περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα θα μας προστατεύσει από την ρωσική απειλή. Δεν το λένε πολύ ξεκάθαρα, αλλά τέλος πάντων αυτό θεωρούν και συνεχίζουν να θεωρούν ότι η Ρωσία είναι ένας αντίπαλος εν δυνάμει που μπορεί να επαναφέρει την, ε, τον ψυχρό πόλεμο. Ε, ασφάλεια και άμυνα πάντως είναι σημαντική και εδώ η Ευρώπη μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στο, στην ασφάλεια μέσα στο μοντέλο που θέλουμε σήμερα είτε μέσα σε συνδυασμό είτε αποχωρισμένα από το ΝΑΤΟ. με τη συμμετοχή των χωρών που θέλουν να το κάνουν. Πρέπει να σας πω ότι προς το παρόν λίγες χώρες ε, ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή άμυνα αυτή καθεαυτή. Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία αλλά λίγες χώρες έχουν πραγματικά ε, δουλέψει για αυτό το τομέα. Για την αλλαγή του κλίματος. Προφανώς θα πρέπει να ξαναρχίσει η συζήτηση, είναι αναπόφευκτο να συνεχιστεί, η συζή, να ανοίξει ξανά η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Δεν ξέρω ποια θα είναι, ποιο θα είναι η έκβαση, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι μιλάμε για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και για τις συνέπειες στο περιβάλλον, για την ασφάλεια και ό,τι θέλετε και ένα από τα βασικά στοιχεία Τη συζήτηση αυτή που θα επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, η πυρηνική ενέργεια δηλαδή, να αποκλείεται από τη συζήτηση. Τρίτο ζήτημα. Με ρωτήσατε το κοινοτικό δίκαιο για τους τομείς που αφορούν τους πολίτες εφαρμόζεται λιγότερο από το κοινοτικό δίκαιο που αφορά πιο οργανωμένες δομές. Αυτό με, με ανησυχεί θα πρέπει να μιλήσουμε με τον Λαμασούρ ακριβώς για το ζήτημα αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα. Σχέση ένωσης και εθνικισμού. Εγώ που συνδέεται με την ταυτότητα. Εγώ πιστεύω πάντα ότι η ταυτότητα έχει περιλαμβάνει το δικαίωμα, τη, την, την, ε, τη συμμετοχή. Αλλά δεν είναι το δικαίωμα, είναι το αίσθημα συμμετοχής. Το αίσθημα το ότι ανήκεις κάπου. Ο εθνικισμός το είπε κάποιος Γάλλος, η, η, ανάδειξη του εθνικισμού είναι να δημιουργείς εκ νέου το παρελθόν για να βγάλεις κάτι από το παρελθόν που δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό δεν πρέπει να το μπεδεύουμε με ένα σύστημα αποκέντρωσης του εθνικού κράτους προς τα κάτω και προς τα άνω. Εφόσον αυτή η αποκέντρωση είναι οργανωμένη. Μία αποκέντρωση προς τα κάτω και προς τα άνω είναι πιο λειτουργική και δεν χάνει τα στοιχεία της εθνικής συνοχής και κατά συνέπεια τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν προς τα, να κάνουν την αποκέντρωση προς τα άνω ως κάτι πολύ πιο λειτουργικό. Έναντι της μονομερούς συμπεριφοράς δεν μπορούμε να θέσουμε ε, το αντίπαλον δέος της πολυμέρειας χωρίς να υπάρχει μια περιφερειοποίηση οργανωμένη ο, η, η, η καθαρή πολυμέρεια, η πολυμερή, δηλαδή η πολυμερή συμπεριφορά χωρίς συνεργασία δεν οδηγεί πουθενά. Το λέει και η ιστορία αυτό. Τώρα, το θέμα της ε, ιστορίας του καθενός. Ε, υπάρχει μια συζήτηση ακριβώς και για το ρόλο της ιστορίας στα πλαίσια του εθνικισμού ε, που φτάνει μέχρι την περιφέρεια. Το ευρώ. Μπορεί το ευρώ να είναι τοπικό νομίσμα ή παγκόσμιο. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το δολάριο. Το είδαν κάποια στιγμή και οι Κινέζοι όταν ξεκίνησε το ευρώ και πέρασαν τμήμα των αποθεμάτων τους στο ευρώ γιατί πίστευαν ότι αυτό θα ανέβαινε. Η πολιτική γειτονία είναι εξωτερική πολιτική και αυτή, ε, κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας ε, που δεν θα πρέπει να αγνοείται. Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι μοντέλο που μπορεί να το θέλουν και άλλοι, να θέλουν να, το μιμηθούν και άλλοι, με κοσούρ και αλλού. Ε, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να προσφέρουμε στους εξωτερικούς συνομιλητές μας την ε, ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να ε, είναι αντικείμενο μίμησης, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτή την ιδέα της δημιουργίας περιφερειακών ενώσεων, αυτό που λέμε ανοιχτό περιφερισμός, αλλά δεν ταιριάζει παντού αυτό. Η Κίνα είναι μια χώρα με 1,3 δις έχει τη δημογραφική δυνατότητα να γίνει ε, περιφερειακή ε, δύναμη και μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να συνεργαστεί με άλλους κατά ανάγκη. Η αξιολόγηση του κόστους του να μην υιοθετήσουμε μια στρατηγική δράση. Όντως είναι ε, σημαντικό αυτό, αλλά εάν δεν τηρήσουμε τους στόχους μας στην ενέργεια, στη, και αν δεν ε, αναμορφώσουμε την οικονομία μας αυτό θα έχει κόστος και στο κράτος πρόνοιας. Ταυτότητα. Επαναλαμβάνω. Ε, η ταυτότητα είναι κομμάτι της, του αισθήματο. Είχα μια συζήτηση με έναν ε, φιλόσοφο και του είχα πει κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάω με τον Χέλμουτ Κόλ που είναι Γερμανός, αισθάνομαι ε, μια σχέση. Όταν μιλάω με ένα Λατιμο, Λατινοαμερικάνο και ένα Γερμανό, καταλαβαίνω ίσως ότι έχω κάποια κοινά στοιχεία με τον ένα, κάποια κοινά στοιχεία με τον άλλο. Όταν μιλάω όμως με έναν Γερμανό και έναν Ιαπωνέζο, καταλαβαίνω ότι είμαι Ευρωπαίος πολύ εντονότερα. Κάτι παρόμοιο ε, εμφανίζεται και στην συζήτηση ταυτότητα της Ένωσης. Το πρόβλημα της ταυτότητας της Ένωσης είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν λαοί που θέλουν να μετάσχουν σε αυτό το κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν και μπορούν. Και όταν πάψουν να το θέλουν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να πάψουν να ανήκουν. Αλλά το να μετέχεις κόντρα στο κοινό όραμα της Ένωσης είναι κακό για όλους. Και για αυτούς που θέλουν και για αυτούς που δεν θέλουν. Και που μένουν μέσα γιατί είναι υποχρεωμένοι να μένουν. Και αποτελούν το για το κοινό έργο. Το αίσθημα λοιπόν του ανήκειν πρέπει να στηρίζεται σε ένα άθροισμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αποτελούν ένα σύνολο συμπληρωματικής ηθαγένειας. Εγώ βλέπω μερικές, θέλω μερικέ φορές να δω ότι αυτοί που δεν θέλουν να μετέχουν η χώρα του στην Ευρώπη να κερδίσουν τις εκλογές τέλο πάντων και να πάρουν τη χώρα τους και να φύγουν. Να είναι ικανοποιημένοι αυτοί και να είμαστε κι εμεί ικανοποιημένοι που πιστεύουμε ότι είναι καλή η Ευρώπη. πολιτικό μανιφέστο ή πλάνο δράσης, ε, έγινε λόγος για το απρόβλεπτο χαρακτήρα στον κόσμο, μια κρίση μπορεί να θεωρηθεί ως ε, παγκόσμια δικαιοσύνη. Το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι πιο δίκαιο σε σχέση με άλλα μοντέλα. Μπορεί να χρησιμεύσει αυτό. Τώρα, αν η ομάδα θα έπρεπε να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο με ε, λειτουργική ικανότητα, τα θεσμικά είπε κάποιος δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Όντως, για, να, για τον πολίτη, ε, δεν είναι εύκολο να μιλάμε για θεσμικές αλλαγές χωρίς να λέμε γιατί χρειαζόμαστε το μεταρρυθμισμένο ας πούμε θεσμικό όργανο. Αν, αν πούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό χρειαζόμαστε το εργαλείο αυτό, ε, είναι εύκολο να το πούμε. Αν λέμε θέλουμε αυτό το εργαλείο χωρίς να λέμε γιατί το θέλουμε, δύσκολα μπορεί ο πολίτης να καταλάβει. Εγώ όμως θα είμαι πολύ προσεκτικός και θα προσπαθήσω να μην βγω από την εντολή που μου έδωσε το Συμβούλιο. Ο Κάρλος Καρνέρο είπε ότι υπάρχει μια συνταγματική, συντακτική θα έλεγα κρίση. Η Ευρώπη είναι ένας κοινός δημόσιος, ένας ε, καταμερισμένος δημόσιος χώρος. Στο δημόσιο αυτό χώρο υπάρχουν στη στατικά, άλλη ερώτηση ήταν αυτή, Υπάρχουν σοβαρά νομισματικά στοιχεία, σοβαρά οικονομικά στοιχεία, σοβαρά κοινωνικά στοιχεία. Υπάρχει ένα πακέτο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ένα πακέτο ηθαγένειας που δεν υποκαθιστά την αρχική ηθαγένεια κανενός, αλλά που τη συμπληρώνει και δημιουργώντας μόνο αυτό το αίσθημα συμμετοχής, αυτό το αίσθημα του ανήκει που στηρίζεται σε ένα πακέτο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη, δημιουργούμε αυτό το δημόσιο χώρο. Έτσι δημιουργήθηκαν και τα εθνικά το, ο εθνικός πολιτικός χώρος, όχι αλλιώ. Δεν προϋπήρχαν ε, ανέκαθεν, φτιάχτηκαν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό δημόσιο χώρο που δεν υποκαθιστά το, εθνικό πλαίσιο. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να φτάσουμε όπου θέλουμε. Το είδαμε στα προηγούμενα, στα προϋπάρχοντα κάρχη. Ε, τώρα πώς θα προχωρήσουμε ξανά μια ασφαλή Ευρώπη του 2020. Το να προβλέπουμε μια ασφαλή Ευρώπη του 2020 ε, ε, μας οδηγεί στο να προσπαθήσουμε να τη σχεδιάσουμε. Ε, υπήρξε μια ευθεία ερώτηση. Μπορούμε να κάνουμε συμμαχικές σχέσεις, να έχουμε φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και να έχουμε και την αντιπυραυλική ασπίδα για να προστατευτούμε από αυτήν. Ναι, το μαζί σου δεν σημαίνει ότι δουλεύει, ότι πάντα μαζί στη, στον τομέα της άμυνας. Όταν φύγει ένας ε, πύραυλος κάπου θα πέσει. Από κάπου θα φύγει, δεν μας ενδιαφέρει από που θα φύγει, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα πέσει 3.000 χιλιόμετρα από τον Ατλαντικό, ε, ούτε από τον ε, ειρηνικό. Πάντως δεν να πιστεύω ότι αυτά θα μας προστατεύσουν από τα ιρανικά, από τους ιρανικούς πυράβλους. Ταυτότητα τώρα. Η Ευρώπη των κοινών αξιών μπορεί να περιγραφεί. Δεν είναι πρόβλημα να την περιγράψουμε. Συμφωνούμε με μια σειρά αξιών που αποτελούν τμήμα της ταυτότητας αυτής. Για τους πολίτες μίλησα προηγουμένως ευρωπαϊκή δημογραφία συγγνώμη, περιλαμβάνεται στην έκθεση. Θα συμπεριλαμβάνεται τέλο πάντων και θα αποτελέσει τμήμα της σχέση που θα υπάρξει μεταξύ του δημογραφικού αντικτύπου των μεταναστευτικών ροών για την βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης συνοχής και της εγώ από χρόνια υποστηρίζω ότι η συνταξιοδότηση είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση. όταν έχεις ένα δικαίωμα, το ασκείς. Δεν είσαι υποχρεωμένος ωστόσο επειδή έφτασε σε μια συγκεκριμένη ηλικία να σταματήσεις να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Ό,τι και να γίνει με τον Ομπάμα, η Ευρώπη θα πρέπει να θέσει επιτάπητος τις δικές της προτεραιότητες και να προχωρήσει. Δεν εξαρτάται από τον Ομπάμα. Έχουμε μπροστά μας μια έκθεση για το 2020-30, δηλαδή οι περισσότερες προκλήσεις που έχουμε, ενέργεια, έχουν μεν ένα ορίζοντα το 20-30, αλλά αν δεν ξεκινήσουμε από σήμερα, μην σας πω από χτες, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Μιλώντας για ένα σενάριο εν ώψη του 2020, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα μέχρι τότε. Πολλά πράγματα πρέπει να τα ξεκινήσουμε από τώρα για να καλύψουμε τους στόχους σε 15 10-15-20 χρόνια. Κάποιος μίλησε, είπε Πολύ Ευρώπη, πολλά κράτη, πολύ αόρατη χείρ των ε, κυβερνήσεων. Όπου μπαίνει το κράτος κάνει λάθη, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται και η αόρατη χείρ της αγοράς η οποία κάνει λάθη. Η κρίση ήταν κρίση διότι περιμέναμε ότι η αόρατος αυτή χείρ της αγοράς θα τα όλα. Η αγορά δεν έχει πρόβλημα. Οι κυβερνήσεις έχουν πρόβλημα. Δεν δημιουργήθηκε κρίση από τους πολίτες, αλλά τώρα ο πολίτης αγνοεί, ξεχνά ποιοι δημιούργησαν την κρίση και καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση. Κάρλο, μπορούμε να πάμε καλύτερα ή χειρότερα. Στα πακέτα παρέμβαση που έγιναν, που δεν είναι καλά ή κακά, αλλά είναι αναπόφευκτα, είναι αναπόφευκτα για να μην επιδεινωθούν αυτό που, έκανε αυτό που έγινε. Τώρα, η λειτουργία των πακέτων αυτών μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιες αμφιβολίες. Πρέπει να γίνουν γρήγορα. Καλό είναι πάντα να συζητάμε σε 20-30 χρόνια αλλά όχι για να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Μίλησα για την κρίση για το αέριο, για την αντιπυραυλική ασπίδα. Μου είπαν ότι η ομιλία που είχα δεν έχει ήρμο. Το δέχομαι. Μπορεί και να μην είμαι σε θέση να κάνω κάτι πιο βαθύ. Εγώ έκανα αστικό δίκαιο, αλλά όταν ασχολήθηκα με τις υποθήκες, ε, είπε, έλεγε ο καθηγητής μας, αφού δεν έχουμε βάθος, ας έχουμε ε, ζόφο, σκοτάδι. Ε, όσο πιο σκοτεινός ήμουν μπόρεσα να είναι. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τα στοιχεία προσέγγισης με τον πολίτη δεν είναι εύκολα. Η δυνατότητα να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών κλάους. Έχει πολλές διαστάσεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα του Συμβουλίου και των θεσμικών οργάνων εν γέννη, δύσκολα μπορείς να αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη. Καθαρά επικοινωνιακά. Το ψήφισμα του Συμβουλίου που δημιούργησε την ΟΝΕ και χωρίς να υπάρχει το οικονομικό κομμάτι και η οικονομική διακυβέρνηση, το ψήφισμα αυτό του Συμβουλίου τότε ήταν μία μισή σελίδα. Τώρα έχουμε 70 σελίδες ε, δηλώσεις με ε, αισθήματα. Ανησυχεί το Συμβούλιο για αυτό, δεν είναι ικανοποιημένο από εκείνο, χέρι για τούτο. Ο πολίτης αυτό που θέλει δεν είναι να του πω ανησυχώ ή χαίρο, αλλά αυτό θα γίνει έτσι, εκείνο θα γίνει αλλιώς. Γιατί όλοι πάμε και πίνουμε ε, ένα ποτηράκι και είμαστε ευχαριστημένοι. Η επικοινωνία πρέπει να αλλάξει. Ακόμα και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Για να κερδίσουμε τον πολίτη. Αυτό που είπε ο Λαμασούρ όμως με εντυπωσιάζει πολύ. Το να κάνουμε τους νόμους για τους πολίτες πιο ουσιαστικούς, πιο εφαρμόσιμους. Είναι πολύ καθοριστικό αυτό για να καταλάβει ο πολίτης ότι η Ευρώπη είναι κοντά του. Είμαι σίγουρο ωστόσο ότι οι νέοι που έζησαν σε μια Ευρώπη που δεν εξαφανιστεί το 2020 ούτε το 2030, αν δεν είχαν στη διάθεσή τους τα μέσα που έχουν σήμερα παρά την κρίση στην Ευρώπη, θα εξεγείρονταν. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στην Ευρω... υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο και περισσότερες, ακόμα, ακόμα και αυτές που δεν ήθελαν να μπουν ξέρουν ότι καλύτερα μέσα και ζεστά γιατί έξω είναι πιο κρύα. Ό,τι και να γίνει. Κακή, κάκιστη, αλλά είμαι μέσα. Δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό. Μία χώρα που έφυγε τα 50 χρόνια, τότε θα μου, ε, θα αν μου έλεγε μια χώρα έφυγε τα τελευταία 50 χρόνια, θα έλεγε εντάξει, ξεκινάω η ευρωπαισιοδοξία. Αλλιώ, ε, έτσι και έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φελίπε Μποντζάλες, είδα ότι κρατήσατε πολλές σημειώσεις. Ελπίζω να ήταν καλή η συνάντηση και για σας. Σίγουρα ήταν καλή για μας. Au λοιπόν. So, liebe Kollegen, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. προσγείωση τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης για το, την γενική αναθεώρηση του κανονισμού Richard Corbett εισηγητής ναι ευχαριστώ στην περασμένη συνεδρίαση έκανα μια εισαγωγή στο σχέδιο εκθεσής μου οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω Υπάρχει η ομάδα της Dagmar Roth Beret που έκανε μια έκθεση ήδη. Thank you, Chair. The question has arisen as how we... Λοιπόν, ετέθη το θέμα για το τι θα κάνουμε με αυτή την τρίτη ενδιάμεση έκθεση της ομάδας της Ρότ ε, Μπέρεντ διότι κάποιες από τις ιδέες αυτές απαιτούν για να εφαρμοστούν αλλαγές στον κανονισμό σύγκρουση συμφερόντων μετα... και αρμοδιοτητών μεταξύ επιτροπών, κοινή ε, συνάντηση επιτροπών ε, για να ψηφιστεί μια έκθεση, ε, πολιτική ισορροπία στη σύνθεση των επιτροπών, ψηφίσματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μήπως κάποιες επιτροπές θα πρέπει να γίνουν ειδικέ επιτροπές μήπως κάποιες επιτροπές δεν πρέπει να έχουν πια υποεπιτροπές ή δεν πρέπει να φτιάχνουν ομάδες εργασίας. Βεβαίως όλα αυτά τα θέματα δεν είναι αμφιλεγόμενα. Το να αλλάξουμε τον τίτλο, το όνομα μιας επιτροπής, την κάνουμε ειδική επιτροπή, δεν πειράζει. Αλλά υπάρχουν άλλα θέματα που θέλουν περαιτέρω μελέτη γιατί ε, έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι επί της είναι για λόγους χρονοπρογράμματος. Και για να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα εγώ έφτιαξα ένα σχέδιο κανονισμού που θα ε, απαιτεί το εάν και εφόσον όλες οι προτάσεις της ομάδας εργασίας γίνονται δεκτές από την ε, συνδιάσκεψη των Πρόεδρων. Ε, αυτό το σχέδιο λοιπόν κανονισμού μοιράστηκε αν δεν κάνω λάθος και αν δεν το έχετε μπορείτε κάλλιστα να το πάρετε και να το διαβιβάσετε περαιτέρω. Ε, να μην, τώρα μπορούμε με άλλα λόγια να συνεχίσουμε εμείς τη μελέτη μας ε, χωρίς να περιμένουμε τη διάσκεψη των Πρόεδρων να πάρει απόφαση. Αν μετά ε, εκείνοι αποφασίσουν ότι δέχονται τις προτάσεις, τότε θα πρέπει να δούμε και εμείς αν συμφωνούμε και εμείς και αν πρέπει να αλλάξουμε σε κάτι την έκθεσή μου. Τώρα εγκρίναμε στην περασμένη συνεδρίαση κάποιο χρονοπρόγραμμα. Εγώ λέω τώρα να παρατείνουμε κατά μία εβδομάδα την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Γιατί ε, έτσι θα καλύψουμε και το ενδεχόμενο ε, θα καλύψουμε και την ε, απόφαση αν θέλετε διάσκεψη των Προέδρων αν τηρήσουν αυτή το πρόγραμμά τους. Τώρα, για το αν θα βάλουμε στον κανονισμό μια διάταξη για παρατηρητές στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Παρατηρητές Ε, από εκείνες τις χώρες που αν ίσχυε η συνθήκη της Λισαβόνας θα ήταν ε, υποένταξη κτλ. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ότι κάναμε με την Ανατολική Γερμανία με τους παρατηρητές από εκεί τους δώσαμε δικαίωμα ε, στάτους παρατηρητού στον κανονισμό μας λοιπόν αυτό κάνω εγώ στο σχέδιο κανονισμού που υποβάλλω στην ε, ε, έκθεσή μου. Τώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν θα ήθελα να τα μεταφέρω εδώ για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες κλπ. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν σχετικά φαντάζομαι θα είναι ενδιαφέρουσες και με μεγάλη χαρά θα συναντούσα τις διάφορες ομάδες ή τους συντονιστές των πολιτικών εμάδων για να συζητήσω οτιδήποτε κρεμεί σχετικά με την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ Ρίτσαντ λέει ο πρόεδρος πράγματι θα προτείνω ε, παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου ελπίζοντας ότι έντο μεταξύ θα έχει πάρει την απόφαση της συνδιάσκεψης των Πρόεδρων αν δεν έχουν πάρει την απόφαση τους τι να πω τότε θα πρέπει να παρατείνουμε και πάλι μέχρι τις 19 Μαρτίου ενδεχομένω την ε, προθεσμία αυτή ε, αλλά η 19η Μαρτίου είναι τελευταία ευκαιρία για επιτεύξη συμφωνίας. Προτείνω προς το παρόν τη 10η Φεβρουαρίου ως προθεσμία κατάθεση τροπολογιών εκτός αν πάμε παραπέρα μέχρι το Μάρτιο. Ενρικέ. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστήσω τον Ρίτσαρ ε, Κόρμπετ για την παρέμβασή του. Θα ήθελα να μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την πρόταση εκείνη που έγινε, να βρεθεί τελικά δηλαδή μία λύση που θα μας ε, επιτρέψει να σεβαστούμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας του ε, Κοινοβουλίου και την απόφαση που έχει ληφθεί για τη σχέση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διακυβερνητικής διάσκεψης. Αυτό δεν επηρεάζει τόσο τη χώρα όμως 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία θα αυξηθεί ο αριθμός των μελών εφόσον αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και κατάλαβα ότι είναι μόνο η Γερμανία αυτή η οποία θα χάσει μέλη. Και είχαμε πει ότι ε, θα πρέπει να σεβαστούμε στην περίπτωση εκείνη τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου και ότι αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα τελικά. Αυτό βέβαια εφόσον η συνθήκη της Λισαβόνας το πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Τώρα, έχουμε μία τροπολογία από διάφορες πολιτικές ομάδες, με υποστήριξη από διάφορες πολιτικές ομάδες, όπου λέμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο είχε αποκομίσει μάθημα Γερμανία στην επανένωσή της. Δηλαδή, οι χώρες αυτές που θα βρεθούν με λιγότερα μέλη θα μπορέσουν να προσθέσουν στα μέλη τους και τους παρατηρητές που δικαιούνται και στη συνέχεια τα άτομα αυτά, από τη στιγμή θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη, θα γίνουν πλήρη μέλη. Ήταν και μια, μάλιστα μια προφορική πρόταση που έκανε ο Σαρκοζή στην Αλομέλεια του Δεκεμβρίου. Μήπως να υιοθετούσαμε λοιπόν μια τέτοια προσέγγιση. Βέβαια, Ακόμα και οι Ιρλανδοί είχαν πει ότι θα ήταν μια θετική απόφαση. Καταλαβαίνετε όμως ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών και νομίζω ότι η πρόταση αυτή συνάδει με τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Uh, I'm Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στο παρελθόν στις uh, συζητήσεις για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις καταρχάς. Να συγχαρώ τον κύριο Κόρμπετ για την πολύ δύσκολη ουσιαστική και τεχνική αυτή ε, εργασία που κάνει, πολύ σημαντική όμως και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και Πρέπει να σας πω ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική που γίνεται από τον κύριο Κόρπετ γιατί συνδυάζει διάφορα στοιχεία. Πρώτον, έχουμε τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας για το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, έχουμε το ζήτημα της μεταρρύθμισης του Κοινοβουλίου που η ίδια διαδικασία της μεταρρύθμισης του Κοινοβουλίου έχει μέσα της κάποια στοιχεία προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνθήκη της Λισαβόνας και τρίτον υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Θα ήταν καλό πιστεύω, σκόπιμο, και για τον εισηγητή αλλά και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά τα ζητήματα αυτά γιατί διαφορετικά δημιουργείται μια κάποια σύγχυση και μπερδεύουμε αδίκως τα πράγματα και καταλήγουμε σε κάτι σαν Ιρλανδικό καφέ Arliss Coffee που έχουμε μέσα και καφέ και αλκοόλ. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε και τις προθεσμίες, βλέπουμε τώρα ότι έχουμε μια παράταση κατάθεσης τροπολογιών. Αν βέβαια εργαστούμε επεξεργαζόμενοι με συγχωρεί τα ζητήματα αυτά ξεχωριστά θα πρέπει ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε άλλες προθεσμίες. Να δούμε και ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές ε, επιπτώσεις να δούμε τι θα γίνει και με τις διατάξεις αυτές οι οποίες φέρουν ένα αστερίσκο, που θα τεθούν δηλαδή σε ισχύ την πρώτη μέρα μετά την έναρξη εφαρμογή της σχετικής διάταξης της συνθήκης. Αλλά αν απουσιάζει όμως η συνθήκη, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα άρθρα αυτά. Κάποιες πιο συγκεκριμένε ε, τώρα παρατηρήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας, νομίζω ότι οι τεχνικές ε, τροποποιήσεις που έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σωστές, αλλά δεν ασχολούνται με κάποια θέματα στα οποία ενδεχομένως να είχαμε και κάποιες διαδικαστικές επιπτώσεις όπως η νέα διαδικασία της επιτροπολογίας. Εμείς θα πρέπει να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα και εμείς θα πρέπει να δούμε τελικά αν ε, θα έχει αυτό κάποιες επιπτώσεις για τον κανονισμό μας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να δούμε ή και σε άλλους ε, τομείς. Το ότι το συζητάμε αυτό τώρα και όχι όταν θα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μας αφήνει ενδεχομένως να λάβουμε υπόψη προτάσεις που έχουν γίνει από άλλους συναδέλφους μας, όπως ο κύριος Μασούρ που έχει κάνει κάποιες προτάσεις για την έκθεση Μπρόκ, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Φοβάμαι λοιπόν ότι ε, χάνουμε κατά κάποιο τρόπο την πολύ θετική συμβολή που θα μπορούσαμε να έχαμε από άλλες ε, συναφείς ε, εκθέσεις που ασχολούνται και αυτές με τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις επιπτώσεις της εφαρμογής συνθήκης αυτής. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο και να περάσουν τα στοιχεία αυτά και στις, ε, να λάβουμε μάλλον τα στοιχεία που έχουμε από τις ε, εκθέσεις διάμεσης αξιολόγησης. Τώρα, αναφερθήκαμε και στη διάσκεψη των Προέδρων, η οποία ακόμα συζητά ορισμένα ζητήματα, δεν έχει καταλήξει όμως σε οριστική απόφαση. και όσον αφορά τον ε, κώδικα συμπεριφοράς και τη διαδικασία όσον αφορά τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, το κείμενο νομίζω πηγαίνει πιο πέρα από αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στην ε, ομάδα μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά επισημοποιεί την ε, διαδικασία του να δοθεί εντολή σε αυτόν ο οποίος ξεκινά διαπραγματεύσεις με ένα άλλο θεσμικό όργανο. Νομίζω ότι αυτό υπερβαίνει κάπως την αρχική μας ε, συμφωνία και νομίζω ότι θα πρέπει να καθορίσουμε καλύτερα την όλη διαδικασία συμφωνίας ε, σε πρώτη ανάγνωση και να υπάρχει μια συγκεκριμένη εντολή που να δείτε σε αυτόν ο οποίος ε, διαπραγματεύεται σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν θα πρέπει στη φάση αυτή να επισημοποιηθεί η διαδικασία αυτή του, του να δίνεται δηλαδή εντολή ε, σε κάποιον να διαπραγματεύεται με άλλα θεσμικά όργανα σε πρώτη ανάγνωση. Να το εξετάσουμε λοιπόν περαιτέρω αυτό. Επίσης, ε, πάλι η ομάδα μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προτείνει πολλά περαιτέρω πράγματα όσον αφορά τον ρόλο των συντονιστών αλλά ακόμα πολλές φορές και των ε, σχεδόν εισηγητών και τη δικασία που προβλέπεται στη συνεργασία μεταξύ αυτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα όσα έχει προτείνει για τον ρόλο των συντονιστών η ε, ομάδα μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή ή να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τη στιγμή που δεν μας εθέσει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις γενικότερα αργότερα για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις έχουν ήδη πάρει τις αποφάσεις τους ε, για, το για μετά τη συνθήκη το Δεκέμβριο πάρθηκαν πολλές αποφάσεις και γι' αυτό το, είναι θεμητό και το Κοινοβούλιο να πάρει θέση σχετικά με το τι θα γίνει όταν θα ε, ε, εφαρμοστεί η συνθήκη. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ε, όταν εφαρμοστεί η συνθήκη, αν εφαρμοστεί αν θέλετε. Το... Ε, το πώς θα αντιδράσει η κοινή γνώμη στην Ιρλανδία και κατά πόσο μπορούμε να την επηρεάσουμε προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση είναι άλλος λογαριασμός αλλά νομίζω ότι σε... Ε, τώρα πρέπει να κάνουμε τις σχετικές συζητήσεις που για το θέμα αυτό διότι το καινούριο κοινοβούλιο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχει νόημα να κάνει τις συζητήσεις αυτές θα είναι πολύ αργά τότε. Άρα λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε και Εντάξει δεν λέω θα δούμε το φθινόπωρο τι θα γίνει ε, με την συνθήκη. Ο κύριος Λένε, πρόεδρε, ε, κοίταξα όλες τις τροπολογίες που υπευλήφθησαν. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση είναι αρκετά ισορροπημένη ε, και καλή. Ωστόσο έχω κάποιες παρατηρήσεις. Από μια μεριά ο ρόλος των ε, συντονιστών των επιτροπών ε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές εκεί, που, ε, ε, δεν είναι μη εγγεγραμμένοι έχουν ειδικέ διατάξεις και δικαίως διότι δεν ανήκουν σε κάποια πολιτική ομάδα. η, το χαρακτηριστικό του μη εγγεγραμμένου που δεν ανήκει δηλαδή σε κάποια πολιτική ομάδα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επενέσουμε αν θέλετε ή θα πρέπει να για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα η, η, η πολιτική ομάδα είναι μια ομάδα ατόμων που έχουν τις ίδιες απόψεις και όπου ε, κάποιος από μια πολιτική ομάδα υποστηρίζεται από όλους τους υπόλοιπους λοιπά, Γι' αυτό υπάρχουν και πολιτικές ομάδες. Λοιπόν, ενώ μη εγγεγραμμένος δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, επόμενο θέμα ε, αυτά, ε, ε ευελιξία ε, όπως είπε και ο συνάδελφος Σάιερ ε, στον κανονισμό αυτά τα οποία θα αυτά που θα βάλουμε στον κανονισμό που θα βάλουμε στον, κανό, στον κώδικα δεοντολογία, στον κώδικα συμπεριφοράς ε, αυτά που συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη νομοθεσία αυτά όλα θα πρέπει να τα βάλουμε ε, στον κανονισμό ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει με όλα αυτά να συμβαδίζουν αυτά που λέμε θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα κάτι τι άλλο. Ο πρόεδρος ανέφερε πολλά προβλήματα ε, τα οποία θα μπορούσαμε όμως να ξεπεράσουμε ε, χωρίς να κουβεντιάσουμε ε, το ενδεχόμενο και το να κάνουμε ε, να προσπαθούμε να φανταστούμε ε, τα αποτελέσματα του ενός Ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Εγώ νομίζω ότι με τεχνικές αποφάσεις της Επιτροπής αυτής μπορούμε να προετοιμάσουμε πολλά πράγματα και έχω και αποφύγουμε βεβαίως να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από το τέλος της θητείας, πριν από τις εκλογές ή πριν από το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Αν όμως έχουμε πάρει τις τεχνικές αποφάσεις θα μπορούμε κάλλιστα να αντιστασμοποιήσουμε, να τις επισημοποιήσουμε μετά τις ε, εκλογές το, στην επόμενη θητεία αυτή η ελαστικότητα νομίζω πρέπει να υπάρχει. Τώρα για την... Α, θα πρέπει κάπου να εφαρμοστεί μια διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, μέσα σε αυτό το όργανο και δεν μιλάμε μόνο για το δεν μιλάμε για τον μιλάμε για σοβαρές αποφάσεις αυτή τη στιγμή οπότε τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και θα πρέπει να τα δούμε τώρα για την τροπολογία 82 για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με τον κανονισμό χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο από τεχνικής απόψεως για το μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε βέβαια το Συμβούλιο αλλά γιατί από τώρα θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση σχετικά αν το δούμε το θέμα με το Συμβούλιο ε, και πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα στον κανονισμό, θα αλλάξουμε αργότερα. Τώρα για το τροπολογία 70 για τις ε, ε, χωριστές ψηφοφορίες. Άμα εγώ νομίζω ότι το αίτημα για χωριστές ψηφοφορίες θα πρέπει να προέρχεται από την πολιτική ομάδα και όχι από τις επιτροπές θα πρέπει να ανατεθεί το θέμα αυτό στην πολιτική ομάδα και θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα όριο να πούμε maximum τρεις ε, χωριστές ανά ομάδα. Αυτό όμως δημιουργεί μια ανισότητα γιατί έχουμε μεγάλες ομάδες και μικρές ομάδες. Έτσι και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε αυτό το κατά πόσον αυτό το ανώτατο όριο 3 ή τέλο πάντων αυτή η ιστορία με το 3 είναι σωστή όχι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι προσωπικές μου παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι σε γενικέ γραμμέ είναι πολύ καλά αυτά που προτείνονται εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε, συμφωνώ καταρχάς ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του Κοινοβουλίου σήμερα για να προετοιμάσει την μεταρρύθμιση των διαδικασιών εν ώψη της θέσεως σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να επιβάλλουμε την ευθύνη προσαρμογής των κανόνων του Κοινοβουλίου σε ένα νεοκλεγέν κοινοβούλιο, ιδίως για μια καινούργια συνθήκη. Οι προετοιμασίες λοιπόν για τις αλλαγές που ελπίζουμε ότι θα αναλάβουμε πρέπει να κλείσουν πριν λήξει η θητεία του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να εκθέσουμε εαυτούς στην απειλή να μας μεμφθούν γιατί δεν επιτρέπουμε τη λειτουργία της συνθήκης μόλις τεθεί σε ισχύ. Δεύτερον, πιστεύω ότι η έκθεση Ντεάν που δεν συζητήσαμε ακόμα παρέχει κάποια θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στον κανονισμό ιδίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό της του πρόεδρου της Επιτροπής, συμφωνώ εδώ απόλυτα, με τον κύριο Λένε. Τρίτον, πρώτη ανάγνωση. Η λύση, η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας στην απόφαση σε πρώτη ανάγνωση έγινε πολύ της μόδας. Δεν μπορώ να καταλαβώ. Γιατί πιστεύω ότι στο προηγούμενο κοινοβούλιο 25% περίπου των αποφάσεων συναπόφασης έκλειναν στην πρώτη ανάγνωση. 50 25% στη δεύτερη και άλλο 25% στην τρίτη. Με το τωρινό κοινοβούλιο τα ποσοστά άλλαξαν. 50% των αποφάσεων με συναπόφαση πέρασαν στην πρώτη ανάγνωση, ολοκληρώθηκαν στην πρώτη ανάγνωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε προσεκτικά τις διαδικασίες αυτές και τον κώδικα διοντολογίας ιδίως στον άτυπο τρίλογο που βγήκε από την ομίχλη του. Και να ενισχύσουμε την λειτουργία των σκιωδών εισηγητών από τις ομάδες που δεν έχουν τον επί της ουσίας εισηγητή. Επίσης θα πρέπει να, δούμε μια, έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για τις διαδικασίες ανάθεσης εκθέσεων στην Επιτροπή, στις Επιτροπές, σε μια διαβούλευση που είχα στην ομάδα μου κατακρίθηκε ιδιαίτερη εφαρμογή του, τώρα του άρθρου 45 παραγραφος 2 και του γεγονότος ότι πολλές από τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας πέρασαν από την Ολομέλεια ε, με όχι ικανοποιητικό τρόπο. Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει να ξανασκεφτούμε την αποτελεσματικότητα του άρθρου 45.2 και θα υποβάλω μια σχετική πρόταση. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα Είμαι ικανοποιημένο με την ημερομηνία της 10ης Δευτέρου. Λειτουργική και χρήσιμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ για την έκθεση αυτή. Τώρα, όσον αφορά τη διάσκεψη των Προέδρων και τις αποφάσεις που έχει πάρει η διάσκεψη αυτή, νομίζω ότι ε, όλοι συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αμέσως τα όσα έχουν αποφασιστεί στη διάσκεψη αυτή. Τώρα, τρία ακόμα πράγματα στα οποία θέλω να αναφερθώ. Είναι λογικό να ασχολούμεθα με την συνθήκη της Λισαβόνας. Βέβαια, η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει ακόμα εγκριθεί, πάντως πιστεύω ότι όταν και εφόσον η συνθήκη της Λισαβόνας εγκριθεί θα είμαστε εμείς σε θέση γρήγορα και εύκολα να εφαρμόσουμε τις διατάξεις που συνδέονται με αυτήν και που ενδεχομένως θα τροποποιούν τον καονισμό. Και κάτι τελευταίο το οποίο το συζήτησα πολύ με τον συζητητή αλλά και με άλλους είναι ότι ο κανονισμός θα πρέπει να είναι καταρχάς ένα μέσο το οποίο θα βοηθά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να διευκολύνει ουσιαστικά το έργο μας. Θα πρέπει να ε, εδραιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και όχι να λειτουργεί ουσιαστικά ενάντια στο έργο των Ευρωβουλευτών και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές τροποποίησεις που έχουν να κάνουν με ξεχωριστές ψηφοφορίες και αφαιρούν τελικά δικαιώματα από τους βουλευτές. Αφαιρούν δικαιώματα τελικά από τους ε, ίδιους τους νομοθέτες. Ξέρετε ότι ε, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές οι ξεχωριστές ψηφοφορίες ε, με ύποπτους τρόπους στο παρελθόν, προκειμένου να τροποποιήσουν δηλαδή τη στάση ενός βουλευτή. Καταλαβαίνετε όμως ότι ε, το δικαίωμα για τη ξεχωριστή ψηφοφορία θα πρέπει να ισχύει και ακόμα και αν καταλήξουμε σε χιλιάδες ξεχωριστές ψηφοφορίες νομίζω ότι θα πρέπει το δικαίωμα αυτό να υπάρχει, μέχρι ίσως να κουραστούμε να χρησιμοποιούμε πια τη μέθοδο αυτή. Και ο λόγος για τον οποίο χρονοτριβούμε αυτή τη στιγμή είναι για το ότι οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τα πορίσματα της ομάδας εργασίας για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, ομάδα μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τη Λισαβόνα μπορούν να εξεταστούν αργότερα. Αυτά τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, ας αντιμετωπίσουμε το αστομότερο δυνατό. Δεν ξέρω αν ο Ρίτσαρντ Κόρμπετ θέλει να πει κάτι ακόμη. Εγώ ε, επαναλαμβάνω ίσως κάτι που έχω πει ότι για όλες τις συνθήκες Μάστριχτ, Άμστερνταμ και τα λοιπά ε, υπήρξε προετοιμασία αρχές του 2008 βέβαια μετά την ε, σύνοδο κορυφής της ε, Λισαβόνας ε, ξεκίνησε μια κάποια προ, προετοιμασία αν θέλετε και φτιάχτηκαν αυτές οι, οι προπαρασκευαστικές εκθέσεις αλλά εντωμεταξύ ε, λόγω των ε, μη κυρώσεων ή των κυρώσεων τα πράγματα άλλαξαν μέχρι το, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τι μας είπε, μας είπε ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει τελειώσει και η τελευταία κύριε, κύριος και επικύρωση άρα ε, εκεί μέχρι τότε κάτι πρέπει να έχουμε κάνει. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζονται. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, προετοιμάζεται. Η διάσκεψη των Προέδρων μας έδωσε το πράσινο φως για αυτή τη δουλειά. Γιατί λοιπόν εμείς λέμε όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το μαστιγωνόμαστε και... Ε, και αυτοπεριοριζόμαστε τελικά. Ρίτσαρντ Κόρμπετ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά, για τα καλά λόγια που είπατε για τη δουλειά που έκανα. Βεβαίω ε, ευχαριστής και έπαινε ανήκουν και στη γραμματεία. Βεβαίω το μεγάλο πρόβλημα είναι το χρονοπρόγραμμα και κατά πόσο η έκθεση αυτή πρέπει να χωριστεί στα δυο μετά από αυτά που είπε στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι συντονιστέ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα ή την πιο προηγούμενη τέλο πάντων στο Στρασβούργο για να συζητήσουν ακριβώ αυτά τα πράγματα, να δουν τι είναι ακόμη εφικτό του τελευταίου μήνε ζωή του εδώ του Κοινοβουλίου. Το πρώτο πράγμα που αποφασίστηκε ήταν ότι πρέπει να παραταθούν οι προθεσμίες για την κατάθεση των τροπολογιών και να αναβληθούν ε, ε, για αργότερα οι ημερομηνείς ψήφισης ψηφοφορίας στις διάφορες επιτροπές. Τώρα, για το κατά πόσον θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμεθα με τη συνθήκη της Λισαβόνας όλοι οι συντονιστές εκείνη τη συνάντηση συμφώνησαν ομόφωνα ότι θα ήταν δύσκολο να πάψουμε να ασχολούμεθα με το θέμα αυτό αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να, δουλέψουμε, να δουλεύουμε έχοντας όμως υπόψη ότι τώρα δεν μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές πριν από την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα μπορούμε να αποφασίσουμε αλλαγές μόνο οι οποίες θα άρχιζαν να εφαρμόζονται μόνο μετά την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δηλαδή, οποιασδήποτε αλλαγέ συζητούνται και αποφασίζονται τώρα δεν μπαίνουν στον κανονισμό τώρα. Θα μπουν στον κανονισμό αργότερα. Γιατί πρέπει να αποφασιστούν τώρα. Επειδή ένα από τα πιθανά σενάρια είναι να, γίνει κι άλλο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία στις αρχές του φθινοπόρου η Ιρλανδία θα τα αποφασίσει αυτό. Όμως αν γίνει το δημοψήφισμα και αν οι Ιρλανδοί ψηφίσουν ναι, τότε η συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί σε ισχύ τέλος του 2009, αρχές του 2010, αλλά πιθανόν και 1η Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου του 2009 αν γίνει κάτι τέτοιο, το καινούριο κοινοβούλιο που θα έχει βγει από τι ευρωεκλογέ δεν θα έχει το χρόνο να τα κουβεντιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Ο κύριο Λένε Θαρό είπε ότι θα μπορούσαν να παρθούν κάποιε αποφάσει τώρα στην Επιτροπή και μετά το καινούριο κοινοβούλιο να πάρει την επίσημη απόφαση. Όχι, ε, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται αυτό. Και βεβαίω, όπω είπε και ο κύριο Νταφ θα έχουμε καινούριου ευρωβουλευτέ που δεν θα ξέρουν τη διαδικασία διαδικασία κτλ. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε επιτυχημένη διαδικασία. Αλλά και αυτό δεν θα έδινε μεγάλο χρόνο. Πάντως κάποια πράγματα πρέπει να ισχύουν, διότι από την πρώτη μέρα θέση ισχύ της νέας συνθήκης τη Λισαβόνας κάποια πράγματα θα πρέπει να αποφασιστούν παραδείγματο χάρη σε σχέση με τη νέα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Α, θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ξέροντας όμως τι παίρνουμε τις αποφάσεις για να τις παρκάρουμε κάπου να τις έχουμε εν αναμονή χωρίς να προδικάζουμε τίποτα για το τι θα γίνει μελλοντικά. Όσον αφορά τώρα την το διαχωρισμό σε δύο διαφορετικές ε, εκθέσεις ή σε παραπάνω από μια έκθεση σε τρεις παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε και οι τρεις, οι δύο οι τρεις εκθέσεις που θα, στις οποίες θα χωριζόταν του εδώ η έκθεση θα πρέπει να ακολουθήσουν όμως το ίδιο χρονοπρόγραμμα έτσι ίδια στιγμή ψηφοφορία, ίδια ολομέλεια κτλ. Πρακτικά δεν, ε, δεν έχει νόημα νομίζω. Λοιπόν, τώρα για το, τροπολογία 4 δεν έχουμε βάλει εκεί αστερίσκο γιατί ε, ε, ε, ήδη οι, ε, δημοσιονομικές προοπτικές έχουν αλλάξει όνομα και ονομάζονται πολιετής κτλ. Αυτό δεν σχετίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα Βεβαίως εγώ λέω να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να έχουμε κάποια πράγματα έτοιμα γιατί σε δίκη της Λισαβόνας όταν αρχίζει να εφαρμόζεται. Αλλά όμως κα, αλλά ίσως θα πρέπει έξι μήνες μετά την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας να αναθεωρήσουμε τα πράγματα, να ξαναδούμε ποια είναι η πείρα που αποκομίσαμε την εφαρμογή αυτών των πραγμάτων και ενδεχομένω να αλλάξουμε πάλι τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα Υπάρχουν αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν ε, προσωρινές ή ενδιάμεσες κτλ. Αλλά όχι αλλαγές ε, του, βασ, του κανονισμού ακόμη ε, και εάν το καινούργιο κοινοβούλιο ε, ζητήσει σε έξι μήνες να αλλάξει ορισμένα πράγματα αυτά δεν είναι η ουσία του κανονισμού τώρα ε, πήγαμε πιο μακριά από αυτά που ζήτησαν οι συντονιστές όχι απλώς είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι φαντάζομαι σε, για ορισμένα θέματα αλλά αν ανησυχείτε για ορισμένα πράγματα είτε τα μας και θα τα δούμε τώρα για τους συντονιστές βέβαια τροπολογία 75 εκεί δεν λέγεται ότι οι μη εγγεγραμμένοι ελέγχουν, συμμετέχουν στην ε, εκλογή, με συγχωρείτε, εκλέγουν τους συντονιστές κτλ. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο, δεν λέμε σχετικό επίσης επειδή ο πρόεδρος μου ζητάει ουσιαστικά να σταματήσω κάποια άλλα θέματα τα αφήσω το κουβεντιάσουμε διμερώς. Α, οι χωριστές ψηφοφορίες δεν αλλάζω τίποτα στα δικαιώματα των ο, ο, μελών να ζητήσουν χωριστή ψηφοφορία. Αυτό που προτείνω εδώ είναι το εξής. Ε, λέω ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία ψηφοφορίας μπορεί να πάρει πολύ μεγάλο χρόνο στην Ολομέλεια λόγου χάρη. Αν λέω λοιπόν ότι αν οι τροπολογίες είναι παραδείγματο χάρη πάνω από 50 ή, ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Επιτροπή σαν φίλτρο. Αν δεν υπάρχει μεγάλη υποστήριξη να μην πάει στην Ολομέλεια η τροπολογία. Γιατί δεν γίνεται αυτό ήδη από τώρα. Ε, όχι μόνο λόγο χωρίς χωριστών ε, χωριστής ψηφοφορίας αλλά και άλλους λόγους αλλά για τις χωριστές ψηφοφορίες θα πρέπει μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με αυτό που περιγράψα προηγούμενα δηλαδή αν δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη για κάποια χωριστή ψηφοφορία να μην ε, ε, ε ταλαιπωρείται ολόκληρη ολομέλεια και ολόκληρο το σώμα ε, με τη χωριστή ψηφοφορία και να χάνουμε το χρόνο μας. Ωραία, 10 Φεβρουαρίου λέει ο πρόεδρος, η προθεσμία πολύ ωραία. Ευχαριστώ Ρίτσαρντ. Πολύ καλή δουλειά έκανες. Και με δύο λόγια τώρα το επόμενο θέμα. Μία έκθεση που έχω κάνει εγώ για τον νέο ρόλο του Κοινοβουλίου, Umbrella Report, δηλαδή μια εργασία που έχει γίνει από όλε τι επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να δούμε τι νέε δυνατότητε που δίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν διαβάσετε την έκθεση, θα δείτε ότι το κοινοβούλιο μας τελικά βγαίνει κερδισμένο από την συνθήκη και η κοινοβουλευτική διάσταση τελικά σε πολύ μεγάλο βαθμό βελτιώνεται και αυξάνεται. νομίζω θα ήταν πολύ καλό να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες από τις ιδέες αυτές στην προεκλογική εκστρατεία. Να ξέρουν δηλαδή και οι ίδιοι πολίτες ότι πάνε να εκλέξουν έναν δυνατό θεσμικό πλεονόργανο, εφόσον βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε εφαρμογή. Μπορείτε λοιπόν να διαβάσετε την έκθεση αυτή και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε αύριο μετά την παρέμβαση της Τσεχικής Προεδρίας ή να αφιερώσουμε τώρα δύο-τρία λεπτά σε παρεμβάσεις, εφόσον θέλετε να πάρετε το λόγο. Διαφορετικά μπορώ να σας πω ότι μπορώ να θέσω την 4η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών. Πρόκειται για μια σφαιρική, όπως σας είπα, συλλογική έκθεση που ουσιαστικά προσπαθεί να παρουσιάσει συλλογικά ποια, πώς θα διαμορφωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη νέα συνθήκη. Θέλει να πάρει κανείς το λόγο. Δεν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς το λόγο λοιπόν. 4 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Θα σας δω αύριο το πρωί στις 9 η ώρα τσεχική ε, προεδρία και μετά σωρό ψηφοφορίες ε, που έχουμε να κάνουμε. Ο πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς.